Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Υπάρχει ένα επιπλέον σημείο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω στην ημερήσια διάταξη. Λάβαμε ένα κατεπήγον αίτημα από πλευράς του κυρίου Γκέρενς, ο οποίος ε, ήταν ο εισηγητής για τα συνοδευτικά μέτρα στον τομέα της μπανάνας ε, και τη συνεργασία στην ανάπτυξη και θέλει να προσθέσουμε στην ημερήσια διάταξη μία ανταλλαγή απόψεων για τη διαδικασία της ε, συνδιαλλαγής μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής φυσικά για το θέμα αυτό και άλλα θέματα ε, στον τομέα της εξωτερικής δράσης, τα οποία αποτελούν αντικείμενο αυτής της συνδιαλλαγής. Η συνδιαλλαγή αυτή ολοκληρώθηκε στις 25 Οκτωβρίου και η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε το ε, κοινό κείμενο στο οποίο κατέληξαν ε, τα θεσμικά όργανα στη διάρκεια 8 τριμερών συνομιλιών που έγιναν μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ως εκπρόσωπος λοιπόν ε, της ε, ομάδας του Κοινοβουλίου στη Συνδιαλλαγή υποστηρίζω προσωπικό στην πρόταση του κ. Γκέρεντς. Δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε να προσθέσουμε το σημείο αυτό στην ημερήσια διάταξη σήμερα και ε, θα συζητήσουμε αμέσως το θέμα αυτό, αμέσως μετά τις ψηφοφορίες. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες ενστάσεις ή κάποια σχόλια για το σχέδιο ημερήσιας διάταξης ως τροποποιήθηκε αν όχι εγκρίνεται. Εγκρίνουμε επίσης και τα ε, πρακτικά της ε, συνεδρίασης της 4ης Οκτωβρίου και της 10ης και 11ης Οκτωβρίου. Τα έχετε λάβει, αν έχετε παρατηρήσεις, ε, σας παρακαλώ να το επισημάνετε στην γραμματεία πριν το πέρας της συνεδρίασης, αλλιώς θα θεωρήσουμε ότι εγκρίνονται. Να δούμε επίσης και τα πρακτικά της 11 Οκτωβρίου του 2011 με τα Εθνικά Κοινοβούλια. Λάβατε τα πρακτικά της κοινή αυτής ε, συνεδρίασης ε, Επιτροπών Ανάπτυξης και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αν έχετε κάτι να επισημάνετε, σας παρακαλώ να το επισημάνετε στη γραμματεία πριν από το τέλος της συνεδρίασης, αλλιώς θεωρούμε ότι και αυτά εγκρίνονται. Τα αποτελέσματα τώρα της συνεδρίασης των ε, συντονιστών της 11 η Οκτωβρίου τα έχετε λάβει επίσης. Αν δεν έχετε σχόλια και για αυτά μέχρι το πέρας της συνεδρίασης εγκρίνονται. Δεν έχουμε λάβει ερωτήσεις ε, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση να σας κάνω εγώ. Και θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον κύριο Ντομένικα ε, ε, Ρώσα που την εκπροσωπεί, αν έχει κάτι να μας ανακοινώσει. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να μιλήσω. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα απλώς ε, να κάνω ένα απολογισμό της κατάστασης για το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων το οποίο θα γίνει την Τρίτη και όπως κάθε έξι μήνες ε, θα έχει και ένα τμήμα αφιερωμένο σε θέματα ανάπτυξης. Το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων έχει σταθεροποιήσει τώρα την ημερήσια διάταξή του. Υπάρχει ένα κοινό θέμα συζήτησης για τη διάσκεψη για την αποτελεσματικότητα της αναπτυξιακής βοήθειας νομίζω ότι από αυτού υπάρχει σύγκληση απόψεων, ε, σε μεγάλο βαθμό μάλιστα. Αυτό καταδεικνύει και η έκθεση και το ψήφισμα το οποίο ενέκριναν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην τελευταία συνοδολομέλεια στο Στρασβούργο. Θα γίνουν επίσης δύο συζητήσεις Ανατολισμού. Ε, μία για τα αποτελέσματα της Πράσινης Βίβλου για το μέλλον της ε, αναπτυξιακής πολιτικής και την ατζέντα για τις αλλαγές και θέλουμε απλώς ενημέρωση από πλευράς κρατών μελών για μια σειρά θεμάτων, κυρίως για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η αναπτυξιακή βοήθεια προκειμένου να υπάρχει ε, μια ανάπτυξη που θα περιλαμβάνει τους πάντες και μια ανθρώπινη ανάπτυξη που θα λαμβάνει υπόψη της τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα βασικά στοιχεία της χρηστής διακυβέρνησης. Θα ε, συζητηθούν επίσης και τα θέματα αυτά ε, προκειμένου να γίνει μια διαφοροποίηση για να λάβουμε υπόψη τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, να ε, Επισημάνουμε δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν αναδιμεομένες χώρες που έχουν αναπτυχθεί περισσότερο και έχουν διαφορετικές ανάγκες από τις αναπτυσσόμενες χώρες. Και επίσης η δεύτερη συζήτηση προσανατολισμού θα επικεντρωθεί στα θέματα βοήθεια στον προπολογισμό. Υπάρχει μια πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ώστε ε, να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή μεταξύ των κρατών μελών από ευρωπαϊκή σκοπιά και επίσης ε, τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται τις ε, εναλλακτικές διόδους που προσφέρει αυτό το αναπτυξιακό μέσο που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί μέχρι τούδε επαρκώς. Θα υπάρξει και μία συζήτηση στη διάρκεια του γεύματος ε, που θα συζητηθούν ε, ε, τα θέματα του κέρατος της Αφρικής μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών Υποθέσεων. Αυτά από πλευράς ανακοινώσεων. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και εγώ. Να περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης ενημέρωση για τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τις πράξεις κατεξουσιοδότηση. Έγιναν 7 συναντήσεις σε τριμερές επίπεδο. Και αυτό που μπορώ να σας πω για αυτές τις τριμερείς συνομιλίες είναι ότι θα ήθελα να αντιστρέψουμε λίγο τον τρόπο με τον οποίο συζητάμε. Αντί να δώσουμε απευθεία το λόγο στον κύριο Γκέρεντ, θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μα κάνει αυτή ε, μία ε, παρουσίαση για τα αποτελέσματα αυτών των τριμερών συνομιλιών και ιδίω τα όσα συζητήθηκαν στον τομέα τη μπανάνα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι στη διαδικασία της συνδιαλλαγής ε, Έχουμε συζήτηση μεταξύ των δύο συνομοθετών, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάνει μία απόπειρα να ε, βοηθήσει ώστε να καταλήξουμε σε κάποιο αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η διαπραγμάτευση αυτή ήταν καρποφόρα, φαίνεται άλλωστε και από το αποτέλεσμα και από τα όσα καταφέραμε να επιτύχουμε. Στην αρχή ήμασταν λίγο οριακά από πλευρά χρόνου, διότι ε, αν δεν είχαμε καταφέρει να καταλήξουμε σε απόφαση πριν από το τέλο του έτου, ε, τα κονδύλια τα οποία είχαν προβλεφθεί στον Ευρωπαϊκό Προπολογισμό προκειμένου να χρηματοδοτήσουμε τα ε, συνοδευτικά μέτρα για την μπανάνα θα χάνονταν και φυσικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε από εκεί και πέρα μια γραμμή προπολογισμού στη διάρκεια της επόμενης ε, διαδικασίας προπολογισμού του 2012. Νομίζω ότι εκατέρωθεν και από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και από πλευρά Συμβουλίου υπήρξε η καλή διάθεση προκειμένου να υπερκεραστούν μια σειρά από στοιχεία τα οποία ίσως θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως πράξεις ε, ε, κατεξουσιοδότηση στη βασική πράξη. Ε, πρόκειται για μια διαδικασία που ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Ε, το 2006 που είχε εγκριθεί το μέτρο αυτό δεν προέβλεπε τα πράξεις κατεξουσιοδότηση. Ήταν κάτι το οποίο εγκρίθηκε μετά από τη Λισαβόνα και δεν υπήρχε δυνατότητα να εισαχθούν πράξεις κατεξουσιοδότηση σε μια αρχική βάση η οποία ήταν τόσο ευρεία. Και έτσι είχαμε ε, τα εκτελεστικά ζητήματα όπως είναι τα θέματα στρατηγικής της κάθε χώρας ε, και χρησιμοποιήθηκαν όλα αυτά προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον τομέα. Ε, πρόκειται για ένα συμβιβασμό ο οποίος πιστεύω ότι θα ικανοποιήσει πλήρως και τις δύο πλευρές και κατά την άποψή μας είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Θεωρώ επίσης ότι αυτό που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η προετοιμασία των μελλοντικών χρηματοδοτικών μέσων, ε, τα όσα θα συζητηθούν ε, για του χρόνου δηλαδή, και του χρόνου θα πρέπει να δημιουργήσουμε μία βασική πράξη που θα μας επιτρέπει να εισαγάγουμε και πράξεις κατεξουσιοδότηση και έτσι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα μπορούν να ε, συζητούν επίσης και να ανταποκρίνονται στις βασικές απαιτήσεις του Κοινοβουλίου, δηλαδή να υπάρχει η ίδια εξουσία στις πράξεις κατά εξουσιοδότηση με το Συμβούλιο. Είναι σαφές ότι ε, στα θέματα της επιτροπολογίας η συνθήκη της Λισαβόνας έχει αλλάξει λίγο τους κανόνες. Έτσι, από πλευράς Κοινοβουλίου υπάρχει μια γνωμοδότηση η οποία θα πρέπει να θεωρείται πλέον ότι βρίσκεται στις εκτελεστικές πράξεις ε, και ε, περιλαμβάνει και τους συνομοθέτες οι οποίοι έχουν να διαδραματίσουν και το δικό τους το ρόλο και θα πρέπει στα νέα νομοθετικό μέσα να υπάρχουν και πράξεις εξουσιοδότηση που θα δίνουν την εξουσία το κοινοβούλιο που έχει δικαίωμα βάσει της συνθήκη της Λισαβόνας να έχει. Δεν έχω τίποτα άλλο να προσθέσω. Νομίζω ότι όλοι είναι σύμφωνοι σε, στα όσα καταλήξαμε στο Στρασβούργο. Νομίζω ότι όλοι έδειξαν ότι έχουν την καλή διάθεση να συμφωνήσουν ε, και υπάρχουν και κάποιοι θεσμικοί και νομικοί περιορισμοί τους οποίους πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τους οποίους με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο θα πρέπει να ε, θυσιάσουμε ίσως και ε, προς το συμφέρον των αναπτυσσόμενων χωρών για να μπορέσουμε να βρούμε μια πιο μακροπρόθεσμα βιώσιμη λύση. Ευχαριστώ. Το Συμβούλιο θέλει να λάβει το λόγο. Δεν ήρθε προς το Συμβουλίου. Καλά. Θα δούμε ε, λόγο στον κύριο Γκέρντ, για να ακούσουμε τι αντιδράσει του. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ απεριόριστα τον κύριο Δελαρόζα και σχεδόν πάντα συμφωνούμε. Και πολλέ φορέ οι όμω όμως αυτή τη φορά νομίζω ότι έχουμε βαθιά διαφωνία μαζί του σε σχέση με το πώ ερμηνεύει τα αποτελέσματα του τριλόγου του τριγωνικού διαλόγου, διότι για να θυμηθούμε τι έγινε είχαμε το βασικό έγγραφο εκεί όπου καλύψαμε την ε, θέσπιση αυτού του νέου χρηματοδοτικού μέσου για την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Άρα δεν κάνουμε σαν το 290 να μην υπήρχε. Και γι' αυτό και στο βασικό έγγραφο είπαμε ότι και είχαμε συμφωνήσει όλοι που ψηφίσαμε αυτή την ρήτρα ούτω ώστε να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την ανάθεση αρμοδιοτήτων σε σχέση με την Κομισιόν όμως παρόλα αυτά δεν αποσπάσαμε για κοιτάξτε πρόκειται για απολυστική αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου. Και γι' αυτό επί μήνες αναρωνόμεθα στο πώς θα ισχύσει το 290 που αφορά αυτές τις αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου. Τι έγινε, με λίγα λόγια. Στη συνδιαλλαγή δεν ήθελε να ακούσει για κατεξοδότηση πράξη στο Συμβούλιο. Οπότε και εμείς προχωρήσαμε στην διαλλαγή για να υπάρξει προσέγγιση των θέσεων. Ο καθένας έδειξε όσο καλή πίστη μπορούσε. Και το κοινοβούλιο και άλλοι. Και είχαμε τρεις φάσεις στη συνδιαλλαγή. Πρώτα-πρώτα προκαταρκτικές διαπραγματεύσεις Εκεί λέγαμε ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε τίποτα, λοιπόν τα χάσουμε όλα. Οπότε για να πετύχουμε είπαμε ότι δεν θα πρέπει να το, το, παρακάνουμε και να περάσουμε σε επόμενη φάση. Γιατί νομίζω ότι και οι τρεις πλευρές είπαμε ότι το συντομότερο πάμε στη δεύτερη φάση για τον ίδιο λόγο. Άρα εκεί πέρα είχαμε την ανάπτυξη των επιχειρημάτων και σας επισύρω την προσοχή και κυρίως της Κομισιόν σε κάτι που θα είναι πολύ σημαντικό. Η εντολή του Συμβουλίου ήταν τέτοια σαν να μην υπήρχε το 290. Και ήθελε το Συμβούλιο να τα θίξει όλα, όλα πλην των κατοξιδότητων πράξεων. Και γι' αυτό και αποφασίστηκε να κάνουμε μια ιδιότυπη διαδικασία. Να πούμε ότι δεν συμφωνούμε σε αυτή τη φάση με τις κατεξουδιώτες πράξεις, αλλά τουλάχιστον είπαμε να προσπαθήσουμε να ισχύσει το πνεύμα αυτών των κατεξουδιώτες πράξεων όσον αφορά τα συνοδευτικά μέτρα. Και είπαμε στην Επιτροπή έχουμε προτάσεις και να μας ενημερώσετε για τις προτεραιότητες σύμφωνα με το έγγραφο και τα σχετικά ποσοστά. Έγινε διάκριση όσον αφορά τα κριτήρια της διάθεσης των πόρων και των προτεραιοτήτων, γιατί τα κριτήρια είναι αντικειμενικά. Ο δε ορισμός αυτής της διάθεσης, ανάλογα με το κριτήριο, είναι αριθμητικού τύπου και όχι με πολιτικές επιλογές. Και η Κομισιόν και το Συμβούλιο συμφώνησαν ότι πρέπει να πληρούνται τα κριτήρια όμως το σημαντικό δεν είναι αυτό το, το σημαντικό είναι εκεί που υπάρχει ε, για τις πολιτικές επιλογές ένα, ένα περιθώριο δηλαδή για την επιλεκτή στρατηγική που είπαμε ότι αφορούν τις προτεραιότητες δηλαδή περιβαλλοντική πολιτική τι θα κάνουμε με ναι, αυτές τις χώρες. Πάμε για αναδιάρθρωση, πάμε για αντικατάσταση της μιας παραγωγής με άλλη και με προκειμένου είπαμε ότι απλώς θα πρέπει να μας πούν ποια είναι η ψαλίδα όσον αφορά αυτά τα ποσοστά. Και νομίζω ότι αυτό το κάναμε και δικαιωθήκαμε. Οπότε επανειλημμένα ζήτησε το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί οριστικά για το 290 το Συμβούλιο. Το 290 είναι άρθρο το οποίο αφορά την ευελιξία και αναδεικνύει αυτό το βασικό κείμενο, βασικό έγγραφο το οποίο βασίζεται στη, στη, στη διάκριση μεταξύ εφαρμοστικών πράξεων, καθαρά εφαρμοστικών πράξεων που αφορούν την επιτροπολογία και από την άλλη μεριά των κατευθυντώτηση πράξεων. Αυτά ισχύανε και πριν την συνήθεια της αγώνας, οπότε είχε λόγο τώρα το Κοινοβούλιο, εάν όμως αφορούσε αυτό αρνητική στάση. Όμως αυτό το οποίο θέλαμε να περάσουμε είναι να δούμε βάσει βάση ποιες διατάξεις τώρα μπορεί να έχει αρμοδίσει το κοινοβούλιο. Είπαμε στην αρχή, πριν τη Λισαβόνα. Ε, υπήρχε με ανασταλτικό αποτέλεσμα εάν έλεγε όχι το κοινοβούλιο. Τώρα δεν ισχύει αυτό. Οι κατεξοδότηση πράξεις βοηθούν σημαντικές πολιτικές του Κοινοβουλίου, σημαντικές αποκλειστικέ του Κοινοβουλίου, γι' αυτό και λέμε ότι πρόκειται για ε, ένα βήμα ω τα πίσω σχέση με αυτό το οποίο είχε προηγουμένω. και τώρα έχουμε το Συμβούλιο και από την την Επιτροπή και κάποιους αρκετούς βουλευτές που έχουν θέσει το περιθώριο τη θέση τη επιτροπή. Ξέρω ότι όλα αυτά είναι πάρα πολύ μπερδεμένα, όμως ε, από την άλλη μεριά είχαμε κάποια επιχειρήματα ε, τα, οποία τα, τα εγκρίνει η Κομισιόν, εγώ όμως δεν, δεν συμφωνώ. Και είπαμε τελικά πήγαμε για μια δέσμια μέτρων, δέσμια αποφάσεων που αφορούσε το ICI, το Erasmus Mundus on a voté sur le package. En ce qui concerne la position du Parlement. Τώρα, για όσον αφορά την τοποθέτηση του Κοινοβουλίου, πρέπει να σας πω ότι η αδυναμία μας να να σπάσουμε το παγέτο μας οδήγησε σε αυτό το πρόβλημα όσον αφορά τις κατηγοριότητες πράξεις. Και υπάρχει τώρα μια μια θέση η οποία είναι υπεκφυγή, δεν κερδίζουμε έτσι. Δηλαδή, αυτό το οποίο είχα πει είναι να δούμε, τι, να δούμε με τι προηγούμενα μπορούμε να κατοχυρώσουμε θέση του Κοινοβουλίου. Ναι, αυτοί είπαν θα ικανοποιηθείτε μεθαύριο, αλλού, αλλού, στον ουρανό. Όχι, όχι, όχι επίγεια, επομένως ανταμοιβή, αλλά στον παράδεισο, έτσι μας είπαν. Όμως, με αυτόν τον τρόπο, είπαμε ότι θα πρέπει εγκαίρως να δούμε τι θα γίνει πριν γίνει, πριν αποφασιστεί ο οικονομικός προγραμματισμός 2013-2020. Οπότε θέλω να μου πείτε τι συνέχεια θα δοθεί στο θέμα των πολιτικών που θα ασκεί το Κοινοβούλιο. Δεν τέλειωσε αυτή η υπόθεση. Πρόκειται να ψηφίσουμε το κάθε μέσο πολιτικής χωριστά. Στην Ολομέλεια, νομίζω στη δεύτερη του Νοεμβρίου και εκεί θα έχω έκθεση ή θα ψηφιστεί, καταψηφιστεί και θέλω να μου πει η Κομισιόν πώς βλέπει τη συνέχεια όσον αφορά επομένω τις θέσεις του Κοινοβουλίου. Αυτή η έκθεση τώρα βγήκε από την διαλήνη και αμεσής με τη δική μου, αυτή που έβαλα στην Ολομέλεια. Και δύο φορές είχε αποσπάσει πάρα πολύ μεγάλη πλειοψηφία ψήφων στην Ολομέλεια. Άρα, πέστε μου, σήμερα να μου πείτε, τι συνέχεια θα δοθεί στην έκθεση. Αλλιώ νομίζω ότι χάνουμε την ώρα μα. Α, και κάτι άλλο τελευταίο. Σα το λέω ξεκάθαρα, το λέω και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή. Δεν κατάφερα μέχρι σήμερα να καταλάβω γιατί. Στα πλαίσια των ίσων όρων συνδιαλλαγής και συναλλαγής θέλουμε σε όλους να παρεμβαίνουν παντού, σε όλους εκτός από το κοινοβούλιο. Κάθε χώρα, ο καθένας. Και αν η συνδιαλλαγή δεν αφορά τι κατεξοδοτήσει πράξει, τότε δεν καταλαβαίνω γιατί αφήνουμε να παρεμβαίνουν τα κράτη-μέλη. Είναι επομένω επίση όλε τα συμβούλια, στα πλαίσια του Συμβουλίου, αλλά αυτό πρέπει να ισχύει και για το Κοινοβούλιο. Αλλιώ, αν πούμε ότι είναι αντιπαραγωγική η ανάμειξη του νομοθέτη, τότε τι γίνεται. Έχουμε ανάμεξη δύο συνομοθετών του Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. στην Επιτροπή. Επομένω, να έχω ένα επιχείρημα που να με πείσει ότι θα πρέπει να επιβαίνουν μόνο τα κρατημέλη και όχι το κοινοβούλιο. Περιμένω να ακούσω τι εντράσει σα. Δεν έχω προτείνει τίποτα σήμερα και δεν ξέρω πώ θα αντιδράσει η Επιτροπή σα. Σε αυτά τα αποτελέσματα τη συνδιαλλαγή. Μπέρμαντ. Υπόθηκε ότι έπρεπε να υποθεί. Ένα πράγμα μόνο θα ήθελα να προσθέσω. Ή μάλλον περισσότερα. Καταρχάς, στις διαπραγματεύσεις αυτές, όσον αφορά το κεφάλαιο για την ανάπτυξη, η αρχή των της ισότητας έχει παραμεληθεί. Πιστεύω ότι το Κοινοβούλιο έχει παραμελήσει. Λοιπόν, έπειτα, πιστεύω πως είναι πολύ σοβαρό το γεγονός ότι σε ένα τόσο σημαντικό θέμα οι συζητήσεις για καταμερισμό των κεφαλαίων είναι συζητήσεις τις οποίες το Κοινοβούλιο δεν θα έχει καμία επιρροή. Εδώ δεν έχουμε να κάνουμε μόνο για εφαρμογή. Οι αποφάσεις είναι και πολιτικής βαρύτητας. Έπειτα, η Επιτροπή μας απομονώθηκε. Δεν βρήκε αλληλεγγύη από καμία άλλη Επιτροπή. Αυτό δεν είναι καλό σημάδι για τις ε, διαπραγματεύσεις των επόμενων δύο ετών όσον αφορά τον προϋπολογισμό. Έχει να κάνει με τη θέση της αναπτυξιακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έπειτα, ίσως είναι εν μέρει και δικό μας λάθος, γιατί κάποιοι από τους διαπραγματευτές μας δυστυχώς δεν μπορούσαν να είναι παρόντες. Όλα αυτά λοιπόν είναι κάποιες από τις ε, αδυναμίες που έχουμε στο ζήτημα της δημοκρατίας. Δεν μπορούσαν να είναι όλοι παρόντες. Αυτό λοιπόν πιστεύω ότι θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στην επιρροή του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω στον κύριο Ντομενικό ότι τα συμφέροντα των αναπτυσσόμενων χωρών δεν θα έπρεπε να παραμεληθούν, δεν θα έπρεπε να παραμεληθούν και να υποφέρουν εξαιτία των αποφάσεων του Συμβουλίου και της Κομισιόν. Είναι πολύ σημαντικό το Κοινοβούλιο να έχει μια ισχυρή θέση όσον αφορά τη χάραξη πολιτικής το 2008 είχαμε το ζήτημα με την ε, πολιτική, τη γεωργική πολιτική και την πολιτική ασφαλείας. Εκεί τονίστηκε ο σημαντικό ρόλο των γυναικών στι αναπτυσσόμενε χώρε και το Κοινοβούλιο ήταν αυτό που πάντα τόνιζε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να εργαστεί ακόμα πιο σκληρά την αντιμετώπιση των ε, συμφωνιών που δεν είναι καλές για τις αναπτυσσόμενες χώρες. Συμφέρει τις αναπτυσσόμενες χώρες να είναι το Ευρωκοινοβούλιο ισχυρό. Και αυτό υπονομεύεται εδώ. Ανησυχώ για το μέλλον και ελπίζω να μπορέσουμε να έρθουμε σε μια συμφωνία για να διασφαλίσουμε την ε, θέση μας. Το λόγο στον εαυτό μου, γιατί δυστυχώς δεν μπορούσα να παραστώ στον ε, τριμερή διάλογο, αλλά σε κάποιε συνδέσει πήγα και γι' αυτό μου φάνηκε ότι είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό το ότι έχουμε γνωμοθετικέ αρμοδιότητε βάσει τις συνθήκε. Όμω προσκρούμε ει αυτή την, ε, την, την, την απόλυτη την αντίσταση από πλευρά κοινοβουλίου από πλευρά Συμβουλίου και Επιτροπής. Δεν θέλουν να εφαρμόσουν στα χρηματοοικονομικά μέτρα και μέσα της κατεδοξιοδότησης πράξης. Και μέσα στην κρίση παραπονιόμαστε για απουσία δημοκρατίας. Ότι δηλαδή λαμβάνονται αποφάσεις ερήμην των λαών. Όμως δεν απονέμονται στο κοινοβούλιο, μάλλον δεν αναγνωρίζονται οι ε, αρμοδιότητες που το απονέμει συνθήκη, το οποίο είναι πάρα πολύ θλιβερό. Και ο, ο βασικός μας διαπραγματευτής έχει μεγάλη πείρα και μεγάλες επιτυχίες. Και επομένως πρέπει να ασκήσει παραπάνω πίεση. Τελικά στεμοχτήκαμε, είμαστε μειοψηφία. Οπότε, ε, διχαστήκαμε στην αρχή, μετά είπαμε να μην πειράξουμε το πακέτο, τον, τη δέσμη των μέτρων και, και πάμε τώρα για, για χωριστή ψηφορία. Αν θα πρέπει να δουλέψει μέσα από την πολιτική του ομάδα μέσο προς μέσο DCI συν υπέρ κατά του, του, του μέσου για τις μπανάνες οπότε εμείς θα, έχουμε μπούσουλα το ότι αν υπάρχει κάποιο μέσο αναπτυξιακό αυτό θα το, το ψηφίζουμε Γιώργης, έχετε το λόγο για να κλείσετε δεν θέλει άλλος από άλλη πτέρυγα του Κοινοβουλίου να λάβει το λόγο. Ρωτάει. Και. Αν είναι ναι, και εγώ συμφωνώ με αυτό το οποίο είπατε. Πώς, εκτός μικροφώνου. Alors nous passons au vote. Non, Monsieur Goerens. Να ολοκληρώσω και να βγάλω συμπεράσματα τώρα είναι πρόημο. Θα ήθελα πραγματικό να γνωρίζω τι σκοπεύουμε να κάνουν οι πολιτικές ομάδες. Ε, είναι σημαντική συζήτηση αυτή. Πρόκειται για κάτι πολύ σημαντικό και εγώ θα σας ερμηνεύσω και τι θα προκύψει από τη διαπραγμάτευση και θα σας ερμηνεύσω και στην Ολομέλεια τι φρονεί η πλειοψηφία της ομάδας. Και μετά ψώμεθα. Να σας πω επίσης ότι στο τελικό στάδιο αποφασίσαμε να ψηφίσουμε το πακέτο. Εγώ απήχα διότι ήθελα να ακολουθήσω την επιθυμία των εκπροσώπων των άλλων επιτροπών ε, του Κοινοβουλίου και πρέπει να σας πω ότι ε, σε αντάλλαγμα δεν μας έλαβαν υπόψη, δεν έλαβαν υπόψη τις επιθυμίες μας και αυτό που δεν αντιλήφθηκαν είναι ότι αυτό που παρασπιζόμαστε εμείς είναι και προς όφελος των θεμάτων που θα μπορούσαν να τους αφορούν ε, το αργότερο το 2013. Για να ολοκληρωθούν λοιπόν οι εργασίες μας θα πρέπει ίσως να γίνει μία ακόμα συνεδρίαση πριν από την Ολομέλεια είτε μία συνεδρίαση τη Ολομέλειας είτε μία συνεδρίαση συντονιστών αλλά θα ήθελα να επισημοποιήσουμε τη θέση μας μεταξύ μας ώστε να μην μας κατηγορήσει κανείς ότι στην Ολομέλεια λέμε άλλα αντί άλλων. Η Πρόεδρος, υπάρχει συμφωνία για την πρόταση του κυρίου Γκέρεντ να γίνει μια επιπλέον συνεδρίαση. Να αναθέσουμε λοιπόν στη γραμματεία να βρει ώρα και τόπο. Να περάσουμε τώρα στις ψηφοφορίες. Έχουμε το σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Την έκθεση της Μισελ Σίφελ για τον ε, δημοσιονομικό έλεγχο της ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχετε όλες τις κάρτες σας για την ψηφοφορία. Donc, tout le monde a sa carte de vote. Έχετε όλες τις κάρτες ψηφοφορίας. Donc, l'amendement... Ωραία. Περιμένουμε λίγο ακόμα. Προφορική τροπολογία υπαριθμών 1. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική, ε, συγγνώμη, τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 2, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4, υπέρ, κατά, αποχές,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 Τροπολογία 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ υπέρ ναι, κατά αποχές εγκρίνεται. Να ψηφίσουμε τώρα το σύνολο της γνωμοδότησης ως τροποποιήθηκε με ηλεκτρονική ψηφοφορία, mm -hmm. άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Κάποιος λείπει. Πέραση ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται ομόφωνα. Η κυρία Κέλλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Στην επόμενη ψηφοφορία για την ε, κατάσταση των γυναικών σε περίοδο πολέμου θα ήθελα να διευκρινίσω ότι η τροπολογία 21 δεν ε, ήταν από την ε, μόνιμη συγκητρία μας για τις γυναίκες. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχει μόνιμη συγκήτρια για θέματα Ένταξη και των γυναικών ε, και τη ισότητα μεταξύ των φίλων είναι η κυρία Κρέτσου και δεν θεωρούμε ότι ε, το αντιμετωπίζουμε με τον κατάλληλο τρόπο. Έχουμε ήδη ε, κάποιον αρμόδιο για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Α. Τροπολογία 1. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται.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 Τροπολογία 10 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 14 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 2 προφορική τροπολογία υπ. 2 υπέρ συγγνώμη η τροπολογία 16 λέει πρόεδρος υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική τροπολογία υπ. 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Να κάνουμε μια επαλήθευση. Η ηλεκτρονική επαλήθευση λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, τροπολογία υπαριθμών 21. Ψήφισαν όλοι. Εγκρίνεται. 14 ψήφοι υπέρ, 8 κατά και 2 εποχές. Προφορική τροπολογία 3. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται τροπολογία 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται να ψηφίσουμε λοιπόν τη γνωμοδότηση ως τροποποιήθηκε άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε ψηφοφορία εγκρίνεται ομόφωνα. Να ψηφίσουμε τώρα τη γνωμοδότηση της κυρίας Λεβίν. Τροπολογία 1, 2 και 3 είναι πανομοιότυπες. Επομένως έχουμε μόνο μία ψηφοφορία υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτονται. Και τώρα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση. Θέλετε παλήθευση. Ωραία. Να επαληθεύσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά την τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε τη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και τώρα ψηφίζουμε τη γνωμοδότηση ηλεκτρονικός. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται 19 ψήφοι υπέρ, 4 κατά. Στη συνέχεια έχουμε τη γνωμοδότηση της κυρίας Τρίφλερ. Τροπολογία 1. Υπέρ. 1 υπέρ κατά αποχέ απορρίπτεται 2 qui est pour qui est contre qui s'abstient υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται amendement 3 qui est pour qui est contre υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το 3 προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. Amendement 5, qui est pour. 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προφορική 2. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. γίνει η ηλεκτρονική παλήθευση. Ψηφίζουμε. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Εγκρίνεται. Οκτώ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Εννέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ήταν και η ψηφορία για το σύνολο νομοδότησης όπως τροποποιήθηκε ψηφίζουμε. Δεν ψήφισαν ακόμη όλοι. Le vote est clos. Donc, adopté 21 voix. sûr. 21 ψήφι. Voilà. Και τώρα έχουμε την έκθεση Γιάν Ζαχράντιλ. Αφορά αυτή την συμφωνία ε, ελευθέρων Α, α, τελειώσαμε, τελειώσαμε με αυτήν. Εξετάσουμε την έκθεση τώρα του κυρίου Ζαχραντήλ που αφορά την εμπορική ανισορροπία μεταξύ εμπορικής, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Εισηγητά, έχετε το λόγο. Κύριε Ζαχραντήλ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω στα τσέχικα. Headphones. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται για μία έκθεση. Αυτή η έκθεση αφορά την ανατησιακή πτυχή της σχέσης με Κίνας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ταυτοποιηθείτε λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ελπίζω ζωγόλοι μου τα ακουστικά τους. Έχετε βρει την γλώσσα, την καμπίνα τέλο πάντων για την γλώσσα που θέλετε και σας ευχαριστώ που δώσατε το λόγο. Ότι για ένα σχέδιο γνωμοδότησης που αφορά την αναπτυξιακή επιτυχή της σχέσης ε και Κίνας. Βασικό θέμα εδώ είναι το να ε, προκαλέσουμε αναθεώρηση των ε, σχέσεων και της παροχής βοηθείας στην Κίνα. Είναι λογικό πάντως κατά τη γνώμη μας να γίνει τέτοια αναθεώρηση. Υπάρχουν πάρα πολύ βάσιμα επιχειρήματα προς τούτο. Γιατί η Κίνα του σήμερα είναι η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο είναι μια χώρα που έχει πετύχει εντυπωσιακή οικονομική ανάπτυξη. Μπόρεσαν να αποτινάξουν το ζυγό της Έχουν σημειώσει πάρα πολύ μεγάλη πρόοδο όσον αφορά την ε, χρήση και ανάπτυξη τεχνολογίας komerční vztahy eh, než vztahy eh, které by platily pro nějakou typickou eh, takzvanou rozvojovou zemi. Άρα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά εκείνα που τη χαρακτηρίζουν αναπτυσσόμενη χώρα. Επομένως, σε αυτό μας το κείμενο καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σταδιακά να εξαλείψει την παραδοσιακή αναπτυξιακή βοήθεια. Να αναπτυχθεί μια συνεργασία και να προχωρήσουμε σε κάποιες ε, καθαρά εμπορικές θέσεις, πιο, πιο εμπορικές θέσεις, σχέσεις. Και για αυτό και εμείς τονίζουμε ότι η, η βοήθεια 2007-2010 ήταν 208 εκατομμύρια ευρώ. Επίσης, Πρέπει να σας πω ότι η Κίνα ίδια δίνει ε, βοήθεια σε άλλες χώρες του κόσμου. Πολλές φορές η ανοσιακή βοήθεια είναι η λεγόμενη συνδεδεμένη βοήθεια Δηλαδή υπάρχουν κάποιες ε, προϋποθέσεις εμπορικές. Αυτοί οι πόρους και προϋποθέσεις ανάπτυξη επομένω. Ε, ψυχική βοήθεια χωρίζεται με αυτόν τον τρόπο και επομένως για όλους αυτούς τους λόγους νομίζω ότι επιβάλλεται να αναθεωρήσουμε τις ε, σχέσεις μας με την Κίνα. Και σεβόμεθα ως εταίρο οικονομικό, εμπορικό. Δεν χρειάζεται να σας εξηγήσω το τι γίνεται τώρα που η Ευρωζώνη περνάει αυτή την κρίση και πόσο έχει ισχυροποιηθεί η Κίνα σαν οικονομικός παράγον. Δεν είναι πως με τίποτα αναπτυσσόμενη χώρα. Είναι μια χώρα που μπορεί η ίδια να χορηγεί οικονομική βοήθεια. Και ήδη έχει αναλάβει νερό ρόλο στην αντιμετώπιση της κρίσης στην Ευρώπη. Επομένως νομίζω ότι ήρθε η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιολογήσει εκ νέου τις σχέσεις με την Κίνα. Για αυτή την ενίσχυση που τους χορηγούμε. Θα πρέπει να οι σχέσεις μας να γίνει πιο εμπορική, θα πρέπει επομένως να θεωρηθεί ότι είμαστε επίσης ώρες. Αυτά είναι τα βασικά του περιεχομένου της ε, εκθεσεώς μου. Πρέπει να ακούσω τις απόψεις σας και τις παρατηρήσεις σας. Και ευχαριστώ να συνεργαστούμε, να δούμε τι θα γίνει με την ε, διατύπωση των τυχών τροπολογιών και τελικά να φτάσουμε σε κάποιον ε, επωφελή συμβιβασμό. Αυτά εισαγωγικά. Περιμένω πώς και πώς να ακούσω τις παρατηρήσει σα. Ευχαριστώ. La parole est à Monsieur Lisek. Ο κύριος Λίσεκ. Thank you very much, Chairman. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω πολωνικά, οπότε κρατήστε τα ακουστικά σας. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική γνωμοδότηση, για ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο δεν είναι σημαντικό μόνο για την Επιτροπή μας, αλλά και για την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου και για όλους τους πολίτες που περνούν από ένα κατάστημα στις Βρυξέλλες, στην Πράγα ή όπου αλλού και αν ζουν και διαπιστώνουν ότι τα πάντα είναι γεμάτα με πουκαμισάκια από την Κίνα, παπούτσια από την Κίνα, αλλά ακόμα και φράουλες και χιλιάδες άλλα κινέζικα προϊόντα ε, που γράφουν πάνω Made in China. Ήθελα να πω λοιπόν στον κύριο Σαχραντήλ ότι θα πρέπει να έχουμε κατά νου το γεγονός ότι η σχέση με την Κίνα θα πρέπει να θεωρείται ε, μια διτή διαδικασία. Όπως σα είπε ο κύριο ε, Σαχραντήλ πρόκειται για μια οικονομία η οποία αναπτύσσεται με αλματώδεις ρυθμούς θα μπορούσε κάλλιστα να θεωρήσει κανείς και δικαίω ότι μέσα σε μερικά χρόνια μια θα είναι η πρώτη οικονομία παγκοσμίω και πρόκειται και για μια οικονομία ε, με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει αρκετές δυσκολίες σε εμπορικό επίπεδο με την Κίνα, διότι δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην αγορά της, δεν υπάρχει διαφάνεια στις μεταξύ μας σχέσεις και υπάρχει και έλλειψη επαρκούς προστασίας σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, για τις χώρες της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης όταν απευθύνονται στην Κίνα. Επιπλέον πρόκειται για μια χώρα στην οποία γίνονται πάρα πολλές εσωτερικές αλλαγές. 200 εκατομμύρια άτομα ζουν κάτω από το κατόφλι της ένδυας. Δηλαδή, κάτω από 1,25 δολάρια την ημέρα. Αυτό είναι το κατόφλι της φτώχειας και υπάρχουν 200 εκατομμύρια άνθρωποι που ζουν κάτω από αυτό το κατόφλι στην Κίνα. Επίσης διαπιστώνουμε ότι έχουν γίνει παρόλα αυτά κάποιες πρόοδοι. Στην Κίνα εδώ και μερικά χρόνια ε, έγινε πρόοδος και καταφέραμε να βγάλουμε κάποια εκατομμύρια ανθρώπων από αυτό το κατόφλι της φτώχειας. Γι' αυτό σας έλεγα ότι πρέπει να γίνει μια διτή διαδικασία. Αφενός θα πρέπει να βελτιωθούν αποτελεσματικά αυτές οι εμπορικές συναλλαγές και να καταφέρουμε να ε, πατάξουμε αυτόν τον προστατευτισμό ο οποίος επικρατεί στην κινέζικη αγορά και ταυτόχρονα θα πρέπει να δούμε πού θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε θέματα ανάπτυξης όπως ε, κάνουμε για παράδειγμα στην περίπτωση της Αφρικής. Στην περίπτωση της Κίνας θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε νέα σημεία. Ε, όπως σας είπα θα πρέπει να είναι αμφίδρομη αυτή η διαδικασία. Αφενός θα πρέπει να βελτιώσουμε τις εμπορικές μας σχέσεις με την Κίνα και αφετέρου θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε αυτή τη νέα ε, τάση οικονομικής ανάπτυξης που διαπιστώνουμε στην Κίνα και η οποία ο στόχο έχει να πατάξει την ένδυα στη χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Για να αλλάξουμε λίγο θα μιλήσω και εγώ Ολλανδικά. Δεν ξέρω αν κάποιοι συνάδελφοι πριν από 1,5 χρόνια ε, ήταν στην κοινοβουλευτική συνέλευση των χωρών ΑΚΕ στην Αγκόλα. Εκεί γινόταν μία διαπραγμάτευση και φτάσαμε σε ένα γήπεδο ποδοσφόρου το οποίο χρησιμοποιήθηκε για το Africa Cup και παρόντες ήταν μόνο οι Κινέζοι. Τα οικοδομικά υλικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του γηπέδου ήταν ε, ε, κινέζικα, οι εργάτες ήταν κινέζοι, αλλά και όλα τα υλικά ήταν κινέζικα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι πρόκειται για βοήθεια σε υποδομές. Το γήπεδο αυτό ήταν σχεδόν ε, ολοκληρωμένο, αλλά δεν υπήρχε καμία προστιθέμενη αξία για την Αγγόλα. Η Επιτροπή Ανάπτυξης λοιπόν θα πρέπει ε, να συντάξει μια γνωμοδότηση για τις σχέσεις μας με την Κίνα ώστε να υποδείξει ε, και την πολιτική της Κίνας, να παρουσιάσει λίγο την πολιτική της Κίνας στις αναπτυσσόμενες χώρες. Στο Κοινοβούλιο ειδικήθηκαν τα θέματα των σπάνιων γεών και άλλων ε, πρώτων υλών το σκεπτικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι πώς μπορούν να φτάσουν σε εμά αυτές οι σπάνιες γέες και οι πρώτες ύλες από την Αφρική και να μην πάνε στη Κίνα. Έχω την εντύπωση όμως ότι η Κίνα, πέραν αυτού του γηπέδου που κατασκεύασε, και ως αντάλλαγμα είχε μία σειρά από παραχωρήσεις από την Αγγόλα. υπάρχει και αυτή η βοήθεια υπό όρους. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να αναφέρουμε στη γνωμοδότηση. Προς το παρόν, στη γνωμοδότηση ε, του συναδέλφου δεν αναφέρονται όλα αυτά τα στοιχεία. Η γνωμοδότηση της ε, Επιτροπής ε, Ήτρε αναφέρεται στις σχέσεις αυτές και θεωρώ ότι είναι και ηθική υποχρέωση δική μας να αναφερθούμε στις σχέσεις μεταξύ Κίνας και άλλων αναπτυσσόμενων χωρών. Συμφωνώ με το συντάκτη της γνωμοδότησης που λέει ότι οι σχέσεις με την Κίνα θα πρέπει να διαφοροποιηθούν σε σχέση με το παρελθόν. Η Κίνα δεν είναι πλέον αναπτυσσόμενη χώρα, είναι πλέον ε, ε, μία εκ των χωρών BRICS, είναι μία αναδυόμενη οικονομία. Ο ρόλος της όμως στην Αφρική είναι αμφισβητήσιμος. Θα παρουσιάσω λοιπόν τροπολογίες προς αυτή την κατεύθυνση και θα ήθελα να θέσω και μία ερώτηση προς το συντάκτη της προμοδότησης. Γιατί δεν υπάρχει αυτή η πτυχή, διότι είναι σημαντικό για μας ως Επιτροπή Ανάπτυξης εδώ. Ευχαριστώ πολύ. Κρατήστε τα ακουστικά σας, θα μιλήσω στη γλώσσα μου. Υπογραμμίσατε μια άποψη, η οποία είναι, ε, μια, ε, έχετε κάνει μια γνωμοδότηση η οποία είναι καλή σε αρκετούς τομείς. Έχω όμως ορισμένα σχόλια. Αυτό που θα έπρεπε να κάνει το Κοινοβούλιο σε σχέση με, στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας θα έχει να κάνει με το αν αυτό το εμπόριο είναι δίκαιο ή όχι και επίση, όσον αφορά τους Κινέζους πολίτε, η παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να είναι δίκαιη και να υποφελούνται όλοι από αυτή. Το εμπόριο είναι στην υπηρεσία των πολιτών. Η μείωση της φτώχειας είναι κάτι στο οποίο πέτυχε η Κίνα υπάρχουν πολύ λιγότεροι άνθρωποι στην Κίνα που ζουν σε φτώχεια. Υπάρχει όμως μεγάλη ανισορροπία ανάμεσα στο πώς αυτή η φτώχεια εξαπλώνεται. Υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην επαρχία και στα αστικά κέντρα. Πιστεύω πως πρέπει να κοιτάξουμε να εξισορροπήσουμε την κατάσταση και πιστεύω πως όλοι συμφωνείτε μαζί μου. Μετά από συζητήσεις με τις, κινεζι... με τις ε, κινέζικες αρχές νομίζω πως πρέπει να ε, εξασφαλίσουμε την... το να μην υπάρχει κάποιο κενό Έγινε λόγος για σπάνιες γιές, για δίκαιη παγκοσμιοποίηση. Δύσκολο να φανταστούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Κίνα να ανταγωνίζονται ποια θα έχει πρόσβαση σε όσο τα δυνατόν περισσότερους πόρους. Σημαντικό είναι να βρούμε τρόπο που να χρησιμοποιούμε βιώσιμα τις πηγές αυτές. Στην Κίνα υπάρχουν ορισμένα γκουλάγ κατά κάποιο τρόπο εργασίας όπου οι εργαζόμενοι αναγκάζονται να δουλέψουν 10 έως 12 ώρες την ημέρα κατά από πολύ δύσκολες συνθήκες σχεδόν χωρίς αμοιβή και τα προϊόντα της εργασίας τους εξάγονται στην Ευρώπη. στον τομέα της ενέργειας και επίσης παράγουν, υπάρχουν εργοστάσεις που παράγουν περούκες. Εγώ δεν νομίζω να χρειαστώ και ελπίζω να μην γελάτε. Ε, ίσως εσείς το βλέπετε αστείο, όμως η παραγωγή και η κατασκευή περούκων είναι εξαναγκαστική εργασία. Παραβιάζει όλες τις ε, συμφωνίες για την εργασία. Και αυτό πρέπει να το εξετάσουμε, διότι όλα τα προϊόντα που καταλήγουν στην Ευρώπη, όλοι για παράδειγμα χαίρονται, μπορούν να αγοράσουν ένα φτηνό κατσαβίδι, ένα σφυρί, ένα τρυπάνι. Εάν δούμε από πού προέρχονται, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Πιστεύω λοιπόν πως στην έκθεση αυτή πρέπει να ξεκαθαριστεί αυτό και εγώ θα συμβάλλω όσο μπορώ για να ξεκαθαρίσω την κατάσταση. Κύριε Γκέρεντς, έχετε το λόγο. Εγώ θα ήθελα κυρία Πρόεδρε να πω υπέρ του κυρίου Ζαχραντήλ ότι σε αυτή την γνωμοδότηση ε, έχουμε θέμα περιορισμού χρόνου, χώρου μάλλον, χώρου, χώρου. Οπότε και γι' αυτό έχουμε τις τροπολογίες και έτσι συμπληρώνουμε αυτά που δεν μπορούσαμε να βάλουμε στο αρχικό κείμενο. Με τίποτα βέβαια δεν θέλουμε ε, να ξαναυπάρξει προστατευτισμός. Βέβαια όπως είναι τα πράγματα τώρα επίσης θα πρέπει να αναθεωρήσουμε την ε, κατάσταση σχέση με την Κίνα. Επίσης τώρα θα πρέπει κάπως να χτενίσουμε τις ε, τροπολογίες για να δούμε τι θα κάνουμε όσον αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και Κίνας. Έχει αντιστραφεί η σχέση με την κρίση. δεν, δεν, δεν είναι ουδέτερη η κατάσταση. Και η ομάδα των 20 ακριβώς αυτό ανέδειξε. Την αντιστροφή της σχέσης Κίνας-Ευρώπης. Έχουμε μόνο κάποιες χώρες που έχουν πρόβλημα με το κρατικό χρέος, το δημόσιο χρέος και καλούν την Κίνα να βοηθήσει και όσον αφορά το Ταμείο Σταθερότητας. Οπότε υπάρχει ορατή, υπαρκτή πίεση από πλευρά Κίνα. Επομένως, ναι, είναι δυνατόν να έχουμε μια χώρα που βοηθεί από την ε, Κίνα. Άρα τι, αυτή η χώρα είναι δυνατόν να συνεχίσει όπως πριν να βοηθάει την Κίνα. Γιατί έχουμε κάποιες χώρες οι οποίες μέχρι σήμερα ήταν κατά της κατάρριξης του εμπάρκου του εμπορίου των ε, όπλων. Τώρα όμως βλέπουμε το αντίθετο αυτό που βρίσκεται προηγουμένως εμείς θέλουμε να κατησχύσει το ευρωπαϊκό πρότυπο οι ευρωπαϊκές αξίες. Και επομένω να δούμε τι θα γίνει όσον αφορά αυτή την ε, το σορευόμενο χρέος το οποίο συνέχεια αυξάνει. Άρα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να δούμε πώς κάτι θα αλλάξει όσον αφορά την Κίνα και όσον αφορά τους εταίρους μας το, τις χώρες BRICS. Επίσης πάρα πολύ ωραία τα λέει ο κύριος ε, Ζαχράντη, εκεί που μας λέει αυτή τη σταδιακή κατάργηση ε, της ενίσχυσης όσον αφορά την πολιτική ανάπτυξης και συνεργασίας. Θα το κάνουμε αυτό, όχι έτσι, θα το κάνουμε στα πλαίσια πολιτικού διαλόγου. Να του πούμε, έχετε τα μέτρα, έχετε τα μέσα να καταπονήσετε τη φτώχεια στη χώρα σας. Και επομένως, εσείς ε, έρχεστε και να μας βοηθήσετε όσον αφορά το χρέος μας. Άρα θα πρέπει να αναδείξουμε αυτές τις πτυχές της έκθεσης, να αναδειχθεί ακριβώς ο, ο ρόλος της, ε, της Κίνας που είναι, έχει ρόλο ανταγωνιστικό της Ευρώπης. Να λοιπόν, ποια είναι τα πραγματικά ζητήματα και πώς σκοτίζονται οι προτεραιότητες μας από αυτές, αυτές τις διαφωνίες μας όσον αφορά τις εξουσιοδότηση πράξεις. Ο κύριος έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συνεχίστε να φοράτε τα ακουστικά σας. Γιατί θα μιλήσω μια γλώσσα που είναι ακόμα πιο σπάνια από τα Ολλανδικά. Θα μιλήσω Σουηδικά. Είναι αφελές ε, αν νομίζετε ότι μπορούμε να απομονώσουμε την Κίνα. Θα ήταν όμως τρομακτικό εάν όσον αφορά την εμπορική πολιτική και άλλους βέβαια τομείς, δεν γινόταν λόγος για σεβασμό στις ατομικές ελευθερίες και στα πολιτικά δικαιώματα. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που μάθαμε από την συζήτησή μας για την Βόρεια Αφρική, όπου η οικονομία είναι ένα τόσο σημαντικό θέμα. Ε, είχαμε να υπογράψουμε συμφωνίες με τη Λιβύη. Στη Λιβύη η οικονομική σταθερότητα είναι πάρα πολύ σημαντική Τώρα όμως έχουμε να κάνουμε με μακροπρόθεσμους στόχους. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι η Κίνα θα συνεχίσει να είναι η τεράστια οικονομία που φαίνεται πως είναι τώρα. Μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα της Κίνας στην Αφρική και ίσως ασχολούμαστε περισσότερο με το τι κάνει η Κίνα παρά με το τι κάνει η Αφρική και τι γίνεται στην Κίνα. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε το εμπόριο με την Κίνα. Μπορούμε όμως να κάνουμε τα στραβά μάτια με το στο γεγονός ότι η Κίνα είναι μια δικτατορία που καταπιέζει τους πολίτες της και η εξαναγκαστική εργασία είναι μέρος ε, της ε, καθημερινής ζωής. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τώρα ο κύριος Λάρς Γκράνβαλτ και ο κύριος Γιάκοψ εκπροσωπούν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. My name is Nils Nils Junger λέγομαι. Θα λάβω το λόγο πριν από το Λάρς. Δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Πέραν του γεγονότος ότι απολαύσαμε την συζήτηση και σημειώνουμε όλα όσα προέκυψαν από αυτήν. Προσβλέπουμε στη συνέχεια της έκθεσης και προς το παρόν απλώς σημειώνω τα όσα άκουσα. Ευχαριστώ. We have no further comments also. Δεν έχουμε και εμείς άλλα σχόλια, λέει ο άλλος πρόσωπος Επιτροπής. Ευχαριστώ. Να σας υπενθυμίσω ότι η προθεσμία για κατάθεση προθε... τροπολογιών είναι η 10η Νοεμβρίου στις 12 το μεσημέρι και να δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Σαχραντήλε, αν το επιθυμεί. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για όλες τα σχόλια. Νομίζω ότι υπάρχει ευρεία συνένεση, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση αποκόμισα εγώ, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε τη σχέση μας με την Κίνα σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας. Νομίζω ότι όλοι επ' αυτού συμφωνούμε. Άκουσα πολύ καλά σχόλια σε κάποια πιο συγκεκριμένα σημεία τα οποία θα πρέπει να τονιστούν και να συμπεριληφθούν στην γνωμοδότησή μου. όπως για παράδειγμα την επιθετική πολιτική της Κίνας σε κάποιες χώρες της Αφρικής, ε, τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της καταναγκαστικής εργασίας. Είμαι στη διάθεσή σας για σχόλια. Κάποιοι από εσά είπατε ήδη ότι θα καταθέσετε τροπολογίες. Νομίζω λοιπόν ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό να καταφέρουμε να έχουμε μια συμβιβαστική γνωμοδότηση που θα είναι αποδεκτή από όλη την Επιτροπή μας. Σας ευχαριστώ και πάλι για τα επικοδομητικά σας σχόλια. Είναι πολύτιμα και περιμένω με ανεπομονησία περισσότερα σχόλια και παρατηρήσεις σας εντός της ε, προθεσμίας που ε, σας ανέφερε η Πρόεδρος. Να περάσουμε τώρα στο σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Θα τώρα την ε, έκθεση πάρα πολύ ενδελεχή του συναδέλφου Νόιζερ και αφορά την ε, πρόσβαση εις τις πηγές ενέργειας ε, μέχρι το 2020. Εδώ πέρα έχουμε πάρα πολλές προκλήσεις ε, ενεργειακές, κλιματικές, οικολογικές, οικονομικές και αμπληξιακές και οπότε και ε, εμείς είχαμε ζητήσει ε, από τις αρμόδιες πέσεις του Κοινοβουλίου να μας κάνουν μια μελέτη για το ζήτημα. Και τώρα έχουμε τους τρεις συν ε, εισηγητάς. Την κυρία Άκη Καρόλα Ντρέμπλοφ είναι ερευνήτρια στο Οικολογικό Ίδρυμα του Βερολίνου. Επίσης ο κύριος Αρνό που είναι ο επικεφαλής του τομέα έρευνας και ενέργειας στο Κέντρο Ευρωπαϊκών Πολιτικών των Βρυξελών και επίσης έχουμε και την κυρία Γκλάντα Λάν που είναι ερευνήτρια στο Chatham House του Λονδίνου. Η τρίτη εκ των συνεισηγητών της ε, μελέτη αυτή δεν μπόρεσε να παραστεί δυστυχώ και το δώσουμε το λόγο στον κύριο Νόιζερ ο οποίος θα μας προσθέσει την ε, έκθεσή του. Παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο αγόρευση γιατί έχετε ζητήσει πάρα πολύ το λόγο. Κύριε Νόζηρο, έχετε το λόγο για πέντε λεπτά και κατόπιν ε, όλοι μαζί οι εμπειρογνώμες θα μιλήσουν για 15 λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την εισαγωγή που κάνατε. Τα σχόλιά σας αφορούν την πρόσβαση στην ενέργεια. Η πρόσβαση στην ενέργεια είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και στο μέλλον θα γίνει ακόμα πιο σημαντικό. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα πρέπει να ενταχθεί στο πλαίσιο των ε, στόχων της χιλιετίας γιατί διαφορετικά θα είναι πολύ δύσκολο να τους επιτύχουμε. Θα ήθελα να κάνω ορισμένα αρχικά προκαταρκτικά σχόλια. Υπάρχουν πάρα πολλοί ΜΚΟ που ασχολούνται με την πρόσβαση στην ενέργεια. Για παράδειγμα, έχουμε την Practical Action, Έχουμε την, ε, το Περιβαλλοντικό Ινστιτούτο της Στοκχόλμης, τα οποία εδώ και πολλά χρόνια ασχολούνται με αυτό και προσπαθούν να δουν πώς ε, γίνεται να διευκολυνθεί η πρόσβαση στην ενέργεια και σε ανθρώπους που ζουν σε αγροτικές περιοχές. Θα ήθελα να σας αναφέρω ένα διεθνές συνέδριο που έγινε στη Στοκχόλμη πριν από λίγες εβδομάδες και όπου τα αποτελέσματα αυτού του συνεδρίου συμπεριλαμβάνονται στην έκθεσή μας. Σύμφωνα με το World Energy Outlook 2012, σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε ενέργεια και 7,2 δισεκατομμύρια ακόμα μαγειρεύουν με βιομάζα. Οι περισσότεροι ζουν σε, στην, ε, σε αγροτικές περιοχές, στην υποσαχάρια Αφρική και στην Ινδία. Με μερικούς ε, συναδέλφους πήγαμε εκεί και ασχοληθήκαμε για παράδειγμα με την Κένια. Το 80% των Κενιατών δεν έχουν πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και 5%, 5 του αγροτικού πληθυσμού έχει πρόσβαση. Η πρόσβαση, δεν υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια ούτε για μαγείρεμα ούτε για θέρμανση. Οι στόχοι της χιλιετίας όσον αφορά την εκπαίδευση τώρα. Ε, σε αυτό έχω να πω ότι χωρίς ενέργεια θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στον τομέα της εκπαίδευσης. Κανένα παιδί δεν μπορεί να ε, μάθει χωρίς φως, χωρίς ρεύμα, δεν μπορεί να κάνει τις ε, δουλειές του στο σχολείο και παρόμοιο, παρόμοια ισχύουν για, την, ε, για τα κέντρα υγείας. Τώρα όσον αφορά το μαγείρεμα με βιομάζα, ε, αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα για το περιβάλλον επιτελείται από ψήλωση των δασών με τη μαγειρική με κάρβουνα. Επίση, ο καπνός που παράγεται είναι πολύ βλαβερός για την υγεία. Ο καπνός αυτός έχει κοστίσει περίπου ένα δισεκατομμύριο θανάτους. Ο ΟΗΕ έχει θέσει μέχρι το 2030 ως στόχο την καθολική πρόσβαση στην ενέργεια και το 2012 θα ανακηρυχθεί έτος ενέργειας. Είναι ένα θέμα που η Επιτροπή μας είναι αρμόδια γι' αυτό. Και στην μελλοντική αναπτυξιακή πολιτική θέλουμε να το θέσουμε ως προτεραιότητα. Οι κύριες, τα κύρια σημεία της έκθεσής μου είναι οι στόχοι του ΟΗΕ για την ε, καθολική πρόσβαση στην ενέργεια μέχρι το 2030, η υποστήριξη αυτών των στόχων και η χάραξη πολιτικής σύμφωνα με αυτούς τους στόχους. προσανατολιζόμαστε σε μικρά αποκεντρωμένα ε, κέντρα ενέργειας έτσι ώστε να μπορούν να έχουν ε, πρόσβαση και άνθρωποι σε αγροτικές περιοχές και σε απομονωμένες περιοχές. Αυτό θα επιτευχθεί κυρίω ανάμεσα στην, ε, ε, σύμφωνα με τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωση και ΑΚΕ και αυτή η δυνατότητα θα μπορεί να ενισχυθεί περισσότερο χρηματικά το 2014. θα πρέπει να εξετάσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες την ε, πρόσβαση στην ενέργεια και το πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει στο έργο αυτό. Η καταπολέμηση του βλαβερού καπνού που παράγεται από την καύση βιομάζας είναι ένα σημαντικός στόχος. Δυστυχώς όμως η πολιτική προς το παρόν δεν ασχολείται με την πρόθεση μικρών αποκεντρωμένων κέντρων ενέργειας και θα έπρεπε η καθολική πρόσβαση ε, στην ενέργεια θα πρέπει να αποτελεί κεντρικό σημείο για το όριο συνήκωση. Και θα ήθελα να τονίσω ότι πρέπει να φροντίσουμε από το 2014 και μετά όταν θα τεθούν οι στόχοι της χιλιετίας να φροντίσουμε να υιοθετηθεί η καθολική πρόσβαση στην ενέργεια σε αυτούς τους στόχους. Έχουμε μία έρευνα πρόσβαση στην ενέργεια Θα ήθελα να σας παρουσιάσω ένα σημείο αυτής της έκθεσης που πιστεύω πως αντιπροσωπεύει τις ε, θέσεις μας. Λέει ότι η έρευνα Σύμφωνα με την έρευνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να προωθήσει την χρήση ε, μικρής κλίμακας παραγωγών ενέργειας έτσι ώστε να μπορεί να πολλαπλασιάσει τα προγράμματά της. Χαίρομαι πάρα πολύ για τα σχόλια των συναδέλφων και πιστεύω ότι η δουλειά που έχει γίνει είναι πάρα πολύ καλή. Merci. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος τώρα στους εμπειρογνώμονές μας. Έχετε ένα τέταρτο στη διάθεσή σας και οι δύο μαζί. Ε, αποφασίστε εσείς πώς θα μοιραστείτε αυτό το χρόνο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ και για την εισαγωγή τον κύριο Νόιζερ. Ε, κύριε Νόιζερ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πολύ που μας δίνετε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε την έκθεσή μας στα πλαίσια της έκθεσης του κύριου Νόιζερ. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα ότι έχουμε πολλού κοινού στόχου και πολλά από τα πράγματα τα οποία αναφέρατε ήδη θα αποτελέσουν αντικείμενο και αυτή τη παρουσίαση. Θα είμαι λοιπόν λακωνικό σε αρκετέ διαφάνειε και σα ευχαριστώ γι' αυτό. Η μελέτη που θα παρουσιάσουμε έχει ετοιμαστεί από τρεις διαφορετικούς οργανισμούς και πέντε συγγραφεί ε, συγγραφείς το, από το Κέντρο Ευρωπαϊκών ε, Πολιτικών Σπουδών. Εγώ είμαι από το Ινστιτούτο στο Βερολίνο και έχουμε και την Κλέιντα Λάν από το Chatham House, η οποία δυστυχώς δεν μπορεί να παραστεί σήμερα. Βεβαίως θα παρουσιάσω και το δικό της κομμάτι της έρευνας. Η παρουσίασή μας θα επικεντρωθεί σε πέντε βασικά σημεία κύρια σημεία που αποτελούν και τη δομή της μελέτης. Έχουμε καταρχάς το πλαίσιο πρόσβαση στην ενέργεια για τις φτωχότερες και αναπτυσσόμενες χώρες με ε, επίκεντρο την Υποσαχάρη Αφρική και την Ινδία. Θα ασχοληθούμε με κάποια από τα προγράμματα, μία εικόνα του τι συμβαίνει, τη δομή τους, το μέγεθός τους ε, και ούτω καθεξής. Θα σας δώσω επίσης κάποια στοιχεία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα πλεονεκτήματα του να έχουμε μικρής κλίμακας ανανεώσιμα προγράμματα σε μεγαλύτερο πλαίσιο, πρόσβαση σε χρηματοδότηση για την ενέργεια στη συνέχεια και θα ολοκληρώσουμε κάποια συμπεράσματα και συστάσεις. Ως προς το πλαίσιο λοιπόν, κάποια από αυτά τα στοιχεία έχουν αναφερθεί και στο παρελθόν, αλλά για να ξεκινήσουμε να σας δώσω έναν ορισμό της πρόσβασης στην ενέργεια, ε, που είναι ο ορισμός που χρησιμοποίησαμε στη μελέτη είναι πρόσβαση σε καθαρή, αξιόπιστη και ε, φθηνή ενέργεια, υπηρεσίες για μαγείρεμα, θέρμανση, φωτισμό, ε, χρήσεις ε, παραγωγικές και επικοινωνίας είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε διάκριση μεταξύ τριών διαφορετικών τομέων όταν συζητάμε θέματα πρόσβαση στην ενέργεια. Καταρχά, τι δικαιούχου θέλουμε να έχουμε ω ομάδα στόχο. Θέλουμε νοικοκυριά, ε, εγκαταστάσει υδροελεκτρική ενέργεια. Επίση, τι πηγέ ενέργεια έχουμε. Ορυκτά καύσιμα, ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, ε, ηλεκτρική ενέργεια. Ε, ενέργεια για μαγείρεμα που αναφέρθηκε προηγουμένως, ε, ε λύσεις δικτύου, λύσεις εκτός δικτύου. Υπάρχουν αρκετές λύσεις και η κάθε μία έχει την εφαρμογή της σε διάφορους τομείς. Και τέλος, τα χαρακτηριστικά της πρόσβασης στην ενέργεια είναι πολύ σημαντικά, διότι δεν αναφερόμαστε μόνο σε ανθρώπους που δεν έχουν πρόσβαση σε ενέργεια και καύσιμα για μαγείρεμα, αλλά αναφερόμαστε και σε ανθρώπους που έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια, για παράδειγμα, αλλά η οποία είναι... Ε, ε, πολύ αναξιόπιστη και αυτό φυσικά παρακολεί και τις ε, βιομηχανικές τους δραστηριότητες. Αναφέρθηκε και το θέμα της παιδείας το να είναι ε, φθηνή η ενέργεια ε, είναι επίσης πολύ σημαντική και το να είναι καθαρή αποτελεί επίσης ε, κάτι στο οποίο επικεντρωνόμαστε. Τώρα, γιατί είναι πολύ σημαντική η πρόσβαση στην ενέργεια. Θα είμαι σύντομο εδώ. Υπάρχουν πολλά σημεία που μας ενδιαφέρουν. Το βασικό είναι ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας δεν μπορούν να επιτευχθούν εάν δεν επικεντρωθούμε σε μεγάλο βαθμό στην πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και σε καθαρά καύσιμα για μαγείρεμα. Αυτά τα στοιχεία τα ανέφερε και ο κύριος Νόιζερ. Ήθελα απλώς να σταθώ σε τρία βασικά στοιχεία. Καταρχάς, το γεγονός ότι 1,3 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή περίπου το 20% του παγκόσμιου πληθυσμού, δεν έχουν ακόμα πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια. Οι περισσότεροι από αυτού, ε, το μεγαλύτερο μερίδιο, το 1,1 δισεκατομμύρια ζουν σε περιοχέ τη υπαίθρου, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα για τι περιοχέ τη υπαίθρου και όπω διαπιστώνεται η υποσαχάρη Αφρική είναι η περιοχή του κόσμου με τη λιγότερη πρόσβαση σε ενέργεια. Ένα ελάχιστο ποσοστό έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια και το παράδειγμα τη Κένια νομίζω ότι αναφέρθηκε και προηγουμένω, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό Μόνο το 20% του πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια εκεί. Τα στοιχεία όλα αυτά αποτελούν τροφή για σκέψη. Τέλος, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να επισημάνουμε και αυτό που είπαμε και προηγουμένως. Ακόμα και σε σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια, δεν είναι αξιόπιστη και πολύ συχνά έχουμε διακοπές ε, ρεύματος. Στην υποσαχάρη Αφρική, για παράδειγμα, υπάρχουν υπολογισμοί που λένε ότι το ε, σύνολο των διακοπών ετησίως είναι ένα διάστημα τριών μηνών εμείς έχουμε 12 μήνες αδιάκοπης παροχής ρεύματος και στην υποσαχάρια Αφρική ζουν 3 μήνες χωρίς ρεύμα. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει και αύξηση σε οικονομικό κόστος μέχρι και 7% του ΑΕΠ ετησίως. Όσον αφορά τώρα τις καθαρές εγκαταστάσεις για μαγείρεμα, ε, είναι αντίστοιχα τα ε, στα αποτελέσματα. 2,7 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρά καύσιμα. Πολλοί χρησιμοποιούν ε, κάρβουνα, ακόμα και φύλλα δέντρων, ε, κόπρανα ζώων και το πρόβλημα είναι κυρίως πρόβλημα της υπαίθρου, αλλά ε, είναι πολύ πιο εκτεταμένο. Και πάλι η Αφρική αποτελεί πολύ προβληματική ζώνη, αλλά και η Ινδία και γενικώ ε, η όλη ε, Δυτική Ασία. Με τις τρέχουσες πολιτικές λοιπόν, η πρόβλεψή μας για την ενέργεια και οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις μας καταδεικνύουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε με την ίδια κατάσταση. Το 2030 θα υπάρχουν ακόμα ένα δισεκατομμύριο άνθρωποι χωρίς ηλεκτρική ενέργεια και 2,7 ε, δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν θα έχουν πρόσβαση σε καθαρές εγκαταστάσεις για μαγείρεμα. Χρειάζονται βελτιώσεις παντού, ε, πέραν της υποσαχάριας Αφρικής ε, που δυστυχώς ε, υπάρχει αύξηση του πληθυσμού και επομένω θα αυξηθεί ο αριθμό των ανθρώπων που δεν θα έχουν πρόσβαση σε καθαρή ενέργεια μέχρι το 2030. Βάσει διαφόρων πηγών, ακαδημαϊκών και μη, η καθολική πρόσβαση στην ενέργεια όμως είναι δυνατή. Εδώ έχουμε μια σύγκριση διαφόρων χωρών, ε, τα ποσοστά ε, παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στα για και πώς αυξήθηκαν ε, αν δείτε τώρα το ανοιχτό γαλάζιο, είναι η Ταϊλάνδη μεταξύ της δεκαετίας του 80 και της δεκαετίας του 90 ε, αυξήθηκε κατακόρυφα η παροχή ενέργειας και υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν αντίστοιχα πολύ μεγάλες βελτιώσεις αν το στοιχείο αυτό αποτελέσει προτεραιότητα για τις κυβερνήσεις. Επομένως η δέσμευση των κυβερνήσεων είναι ε, υψής της σημασία, το είδαμε και για τη Βραζιλία και για την Κίνα. Δεν μπορούν όλες οι χώρες να έχουν ηλεκτρική ενέργεια τόσο γρήγορα όσο η Κίνα. Κατά μέσο όρο έχουμε τρει δεκαετίες ε, μέχρι να φτάσουμε σε υψηλά επίπεδα παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. Το κόστος ε, είναι μεταξύ 36 και 48 δισεκατομμυρίων δολαρίων, όχι ευρώ, είναι λάθος στη διαφάνεια, ετησίως μέχρι το 2030. Το μεγαλύτερο τμήμα θα πρέπει να δοθεί από το δημόσιο τομέα και η ηλεκτροδότηση θα είναι το μεγαλύτερο μερίδιο αυτού του κόστους. Στις αστικές περιοχές η ηλεκτροδότηση είναι μέσω δικτύου, αυτή είναι η φθηνότερη λύση για τις ε, ε, πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές. Στις ε, περιοχές της Υπέθρου ε, προτείνουμε να έχουμε μικρότερα δίκτυα ή καθόλου δίκτυα και θα επικεντρωθούμε σε αυτό. Στις λύσεις εντός δικτύου έχουμε πολύ ισχυρή ορυκτή παρουσία, κυρίως άνθρακα, και έχουμε και στα μικρά δίκτυα ή σε καθόλου δίκτυα έχουμε πάνω από 90% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, τα ίδια περίπου στοιχεία έχουμε και για τι ε, καθαρέ εγκαταστάσει για το μαγείρεμα, αλλά το κόστο είναι χαμηλότερο. Επίση, τι επιπτώσει θα έχουμε σε εκπομπέ φαινομένων διοξιδίου του άνθρακα ε, και φαινομένων αερίου του θερμοκηπίου. Ε, λαμβάνονται υπόψη και άλλα αέρια πέραν του διοξιδίου του άνθρακα και εδώ υποθέτουμε ότι έχουμε και υψηλά επίπεδα υγροποιημένου φυσικού αερίου, δηλαδή μια πηγή που χρησιμοποιεί και παράγει αρκετό διοξίδιο του άνθρακα. Τώρα, Στη δεκαετία του 70 και του 80 επικεντρωθήκαμε σε προγράμματα τα οποία ήθελαν να επεκτείνουν το δίκτυο. Είχαμε αρκετά όμως ε, ποσοστά αποτυχίας ε, λόγω ε, αρκετών λόγων. Το γεγονός ότι δεν ζεσμεύτηκαν αρκετά οι κυβερνήσεις, τα φτωχά νοικοκυριά δεν μπορούσαν να πληρώσουν για την ηλεκτρική ενέργεια και επομένως στα νέα προγράμματα θα πρέπει να επικεντρωθούμε περισσότερο σε ενεργειακές υπηρεσίες και όχι τόσο σε επέκταση του δικτύου. Θα πρέπει να δημιουργήσουμε περαιτέρω δυνατότητε. Ε, να υπάρχουν κατάλληλα μέτρα και επικεντρωνόμαστε εδώ και σε θέματα χρηματοδότησης και τεχνικές κατάρτισης και ε, δημιουργία ρυθμιστικών κανόνων κλπ. Επίσης, προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει όσον ε, αφορά το, το, το, εφαρμόσιμο και την βιωσιμότητα. Επίσης έχουμε τώρα διάφορα έργα και σχέδια τα οποία έχουμε αξιολογήσει και ε, η κατάταξη είναι ανάλογα με μέγεθος, δωρητής, ε, ε, ίδρυμα το οποίο συνεργαζόμαστε και βέβαια γεωγραφικά, περιφερειακά τα κατατάσσουμε. Επίσης έχουμε τρεις μελέτες ε, εδώ, στα πλαίσια αυτή τη ευρύτερη μελέτη, μπορεί να δείτε εδώ πέρα ότι όσο το πλήστον αυτά σχετίζονται με ενισχύσει, με επιδοτήσει, όμω ο εμπορικό παράγοντα γίνεται πιο σημαντικό γιατί πιστεύουμε ότι υπάρχει βούληση να καταβληθεί το αντίτιμο για αυτέ τι υπηρεσίε, ακόμα και από του φτωχότερου. Όπω είπαμε και προηγουμένω, το πιο σημαντικό είναι να μπορέσουμε να έχουμε βιώσιμε και, και αντιγράψιμες ούτως υπήν ε, τέτοιες ε, μορφές έργων και να προσαρμόζονται στις ανάγκες του κάθε τόπου και τώρα η Ιάκη θα μας πει τι πιστεύει για τις ε, βιώσιμες ανανεώσιμες φυγές ενέργειας. Να σας πω τι γίνεται με αυτές τις ενώσιμες ενέργειες και να δούμε πώς μπορούμε να έχουμε μορφές όπως η βιομάζα, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και πρώτα πρώτα υπάρχει βελτίωση για το περιβάλλον και για την ανάπτυξη. Μειώνονται οι εισαγωγέ καυσίμων, κτίθηκαν λιγότερο στην συγκέντρηση της κρίσης και επίσης υπάρχει και επίπτωση θετική στην υγεία. Επίσης οι ενέργειες για είναι καλές και για το περιβάλλον γιατί δεν έχουν βλαπτικές εκπομπές φαινομένου θερμοκηπίου δεν μολύνεται το έδαφος κλπ. Και όπως προαναφέρθηκε έτσι θα έχουμε καλύτερη προσβασιμότητα στην ενέργεια και εδώ βασικά μιλούμε για τις ε, περιοχές της υπαίθρου που δεν έχουν πρόσβαση σε αυτό το δίκτυο. Βασικές τώρα ε, ε προκλήσεις έχουν να κάνουν με το περιβάλλον στην αγορά και να δούμε τι γίνεται στο πρατήριμο, τα μονοπόλια, τι γίνεται τους επενδυτές. Κάποιες χώρες επίσης έχουν συγκεκριμένη τιμολόγηση θεσπίσει. Και αυτό αφορά την τύρφη, και άλλες μορφές ενέργειας. Και εκεί υπάρχει αυτή η δική τιμολόγηση, γιατί πολλέ φορέ όμω αυτό το κάνουν για τις περιοχέ που δεν μπορούν να, να πληρώσουν το κόστο για τι μοντέρες μόρφε ενέργεια. Οπότε, το θέμα είναι τι κάνουν οι δωρητέ, οι μη κυβερνικές οργανώσει ή κάποια φορά μπορεί να κανεί να απλώσει το κόστο ε, σε, σε κάποιο χρονικό, χρονική προοπτική τα άλλα τα πρωί. Είπαμε όμως να δούμε τώρα τι γίνεται με την αγορά που περιβάλλει, που στηρίζει αυτές τι μορφέ ενέργειας. Όχι. Δεν έχουμε, δεν μπορεί να γίνει σωστή συντήρηση γιατί ε, έτσι ο κόσμος δεν μπορεί να έχει την πρόσβαση που απαιτείται. Όσον αφορά αυτές τις τεχνικές εφαρμογές, ξέρω εγώ τις συσκευές, και κάτι άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι οι κοινότητε κάθε φορά θα πρέπει ευθύ εξ αρχή να εμπλέκονται σε κάποια διαδικασία λήψη αποφάσεων. Και επίση θα πρέπει να υπάρχει τέτοιου σώρευση γνώση. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τι κοινότητε αυτέ και κατά δεύτερο λόγο είναι δυνατόν να έχουμε συντήρηση από τοπικού παραγωγού. Επίση, να σα πω κάποια άλλα στοιχεία όσον αφορά νέες πηγέ ενέργειας και νερό. Αν δούμε τα βιοκαύσιμα, την καλλιέργεια βιοκαυσίμων υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές ανάλογα με το είδος που καλλιεργείται. Δεν υπάρχει κάποιο γενικό συμπέρασμα, μπορούμε να εξάγουμε. Όμως η... το νερό μπορούμε να το τακτοποιήσουμε ανάλογα με την ζήτηση. Την παροχή νερού μπορούμε να το τακτοποιήσουμε ανάλογα με την ζήτηση. Η ποιότητα του νερού επηρεάζεται από τη χρήση ε, εντομοκτώνων και ε, παρασιτοκτόνων Έπειτα έχουμε τις επιπτώσεις της υδροηλεκτρικής ενέργειας με την κατασκευή φραγμάτων. Τα φράγματα φιλτράρουν τα στερεά απορρίμματα και παράγουν ενέργεια. Η παραγωγή ενέργειας έχει μεγαλύτερη προτεραιότητα και αυτό μπορεί να επηρεάσει την ε, διαθεσιμότητα του νερού για τον γενικό πληθυσμό. Ευχαριστώ πολύ, Άκε. Θα είμαι σύντομος. Πιστεύω ότι θα μας μένει πολύς χρόνος ακόμα. Ε, λίγα λόγια για τη χρηματοδότηση και μετά τα συμπεράσματα. Είναι εντάξει. Ε, έχετε περάσει το όριο των 15 λεπτών. Θα σας δώσω δύο. Δύο λεπτά όσον αφορά την ενέργεια και την αναπτυξιακή βοήθεια, περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια δαπανώνται κάθε χρόνο για βοήθεια. Είναι περίπλοκο το θέμα, εμπλέκονται πολλοί φορεί. Πιστεύω πως εδώ η λέξη κλειδί είναι η συνοχή και η εναρμόνιση. Αυτό είναι πραγματικά ε, αυτό πρέπει να κάνουμε με την χρηματοδότηση και μόνο 20% της αναπτυξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χειρίζεται από την Κομισιόν. Το υπόλοιπο λοιπόν πρέπει να εναρμονιστεί καλύτερα. Ε, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις ε, δυνατότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το να εναρμονίσουμε τα, το ύψος των ποσών από τα διαφορετικά όργανα. Οι τοπικές λύσεις φαίνεται πως παραμελούνται Γι' αυτό λοιπόν αυτό πρέπει να διορθωθεί και, τα, ε, και οι πόροι αυτοί πρέπει να προσανατολιστούν σε ε, μικρές, μικρές κλίμακας λύσεις, συμπεράσματα. Είναι σημαντική η πολιτική βούληση. Όπως είπα το κανονιστικό πλαίσιο είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχει, ε, δεν υπάρχει one size. Τα έργα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε, της κάθε περίπτωσης. Ε, και, στο τρέινινγκ αλλά και στην ανάπτυξη του έργου. Οι ανανεώσιμες παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο εδώ. Η συστάση μας είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επικεντρωθεί περισσότερο σε λύσεις μικρής κλίμακας και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σε έργα παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις της, ιδιαίτερα εν ώψη του ε, έτους ενέργειας. Και είναι πολύ σημαντικό να μάθουμε, να πάρουμε μαθήματα από τις βέλτιστες πρακτικές, έτσι ώστε να τις χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για άλλα έργα. Ευχαριστώ πολύ και με συγχωρείτε που μίλησα για παραπάνω. Κυρία Κέλλερ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν όντως ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Με χαρά και μεγάλο ενδιαφέρον θα διαβάσω τις έρευνές σας και τις συστάσεις σας. Όσον αφορά την έκθεση του κυρίου Νόιζερ, συμφωνώ και εγώ ότι η έκθεση είναι πάρα πολύ καλή, ότι δεν έχουμε και πολλά να προσθέσουμε ως πράσινοι. Συμφωνούμε με τη γραμμή σας, σε γενικές γραμμές, με την εστίαση στα, στις ανανεώσιμες, με τις αποκεντρωμένες, με τα, τις αποκεντρωμένες ε, πηγές ενέργειας ό,τι πούμε θα είναι συμπληρωματικό αυτόν που εσείς έχετε ήδη αναφέρει στην έκθεσή σας. Επίσης συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία τι ενέργεια χρησιμοποιείται, τι είδος ενέργειας. Αυτό δεν έχει αναφερθεί αρκετά στην έκθεση. Εμείς πιστεύουμε ως πράσινοι ότι οι ανανεώσιμες είναι φυσικά πιο σημαντικές από ότι τα ορυκτά καύσιμα γιατί καταναλώνοντα ορυκτά καύσιμα δεν χειροτερεύει μόνο το ενεργειακό πρόβλημα, αλλά και άλλα, και το περιβαλλοντικό. Και επίση καταστρέφεται το φυσικό περιβάλλον. Ενδεχομένως μάλιστα να, να αναγκάζονται να φεύγουν ε, οι κάτοικοι των περιοχών όπου παράγεται και εξορίζεται ο άνθρακας. Επίσης η καλλιέργεια βιομάζας αποτελεί ενδεχομένως κίνδυνο για την, ε, για την διατροφική παροχή του πληθυσμού. Η ενέργεια θα μας απασχολεί, ελαιόνα και περισσότερο στο μέλλον Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι πραγματικά πρέπει να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο και να το τονίσουμε αυτό στην έκθεσή μας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η περίπτωση της Ταϊλάνδης ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Πώς δηλαδή έγιναν όλα αυτά μέσα σε 10 χρόνια. Και δεν θυμάμαι ποια άλλη χώρα ήταν που αύξησε κατά πολύ το ποσοστά της τελευταία 10, μέσα σε 10 χρόνια. Αυτά για από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Φιάναχολ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, πολύ. πολύ. Μου άρεσε πάρα πολύ η παρουσίασή σας. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και την έκθεση του κυρίου Νόιζερ. Καλύψατε πάρα πολλά και σημαντικά σημεία και δεν έχω και πολλά να προσθέσω. Χαιρετίζω επίσης το γεγονός ότι δώσατε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία του να έχουμε ε, λύσεις εκτός δικτύου ή λύσεις με μικρά δίκτυα και ανεξάρτητες λύσεις και επιπλέον το γεγονός ότι αναφερθήκατε και δύο σε ενεργειακές υπηρεσίες πολλοί από εμά που έχουν βρεθεί σε αναπτυσσόμενες χώρες έχουν βρεθεί στην εξή κατάσταση. Βλέπετε ένα ηλεκτρικό καλώδιο σε μια περιοχή, σε μια κοινότητα, αλλά κανένας δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να έχει πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση και δεν μπορούν να πληρώσουν την ηλεκτρική ενέργεια. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν το γεγονός ότι θα πρέπει να υπάρχουν υπηρεσίες που θα τους επιτρέπουν να έχουν φωτισμό, ε, συσκευές για μαγείρεμα και πρόσβαση σε ηλεκτροδότηση. Δεν αρκεί να υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα που να περνάει από τη γύρω περιοχή. Υπάρχει κάτι ακόμα το οποίο θέλω να αναφέρω και δεν έχει αναφερθεί μέχρι τώρα. Ε, θεωρώ ότι είναι πολύ απαραίτητο να αναφερθούμε λίγο και στην ενεργειακή απόδοση, διότι ιδίως ε, όταν αναφερόμαστε σε μια κοινότητα όπου η παροχή ενέργειας είναι κάπως περιορισμένη έχει μεγάλη σημασία να χρησιμοποιήσουμε στο βέλτιστο δυνατό βαθμό την ενέργεια που μας διατίθεται, ώστε να έχει καλύτερο φωτισμό ε, και περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια με κάθε κιλοβάτ ενέργειας κάποιος. Επίσης, θα πρέπει να εθαρρύνουμε τις αναπτυσσόμενες χώρες να χρησιμοποιούν προϊόντα αποδοτικά ως προς την ενέργεια, όπως κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και, κάνουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες με το Energy Star Scheme, διότι κάθε ε, χωριό θέλει ηλεκτροδότηση που θα χρησιμοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό και αυτό σημαίνει ότι οι επιχειρήσεις ενέργειας δεν θεωρούν ότι είναι δέλεαρ να έχουν μη αποδοτικά προς την ενέργεια προϊόντα σε αυτές τις περιοχές και δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσατε να συμπεριλάβετε και αυτό το στοιχείο στην έκθεση. Ευχαριστώ ο λόγος τώρα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν επιθυμεί να εκφράσει την απόψή τη. Κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ζαν Πολ Ζουλιάν, επικεφαλής του Τμήματος Ενέργειας ε, στην ε, ε, αντίστοιχη Γενική Διεύθυνση. Συμφωνούμε με την ανάλυση του πάνελ και του κυρίου Νόιζερ, ιδίως την πρόσβαση στην ενέργεια στις αναπτυσσόμενες χώρες και θα ήθελα να εμείνω στο γεγονός ότι στην ε, ανακοίνωσή της στην Agenda for Change» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεώρησε ότι η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί προτεραιότητα. Αυτό βέβαια πηγαίνει χέρι-χέρι και με τις προτεραιότητες που καθόρισε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, ο Μπαν Κιμούν, στο πρόγραμμα «Ενέργεια για όλους». Επομένως υπάρχει σχέση μεταξύ ενέργειας και αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε αυτό να το μεταφράσουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, ήδη ασχολείται με θέματα συνεργασίας, αλλά πέραν από τα δυνατότητες πρόσβασης ενέργειας, ασχολούμαστε και με θέματα υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας, ε, θα ήθελα επίσης να αναφέρω ότι η αποκεντρωμένη προσέγγιση την οποία ε, υποστηρίζουν οι εμπειρογνώμονες είναι μια προσέγγιση που υποστηρίζουμε και εμείς. Η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι επίσης αυτό που υποστηρίζουμε και εμείς και είναι σαφές ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν θετικό στοιχείο διότι η αύξηση της κατανόλησης ε, γίνεται με μηδενική επίπτωση στο περιβάλλον δεν έχω περισσότερο χρόνο ίσως, θα ήθελα να εμείνω σε δύο σημεία. Καταρχάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, επικεντρώνεται στην ε, τεχνολογία, αλλά προωθεί ταυτόχρονα και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένες δράσεις όσον αφορά προγράμματα για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Θα πρέπει να είμαστε συνεπείς και ρεαλιστές. 40 δισεκατομμύρια δολάρια όταν τα κονδύλια είναι περίπου το 1 πέμπτο, είναι ε, αυτό το οποίο θα πρέπει να ζητήσουμε από τον ιδιωτικό τομέα και η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα είναι πολύ σημαντική. Θα πρέπει να υπάρχει συμμετοχή και στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και της ενεργειακής απόδυσης που αναφέρθηκε, διότι εμεί θεωρούμε ότι χάνεται ένα 20 με 30% τη ενέργεια στο δίκτυο δυνατοτήτων στι οποίε δεν μπορεί να έχει κανεί πρόσβαση δηλαδή. Θα πρέπει να είμαστε λοιπόν πολύ ε, καλά επικεντρωμένοι και μα ενδιαφέρει και η χρήση του άνθρακα. Στι χώρε ε, της Αφρικής υπάρχουν και μεγάλε δυνατότητε υδροελεκτρική ενέργεια που δεν τι έχουμε εκμεταλλευτεί επαρκώς και πρόκειται για μια πηγή ενέργεια ε, η οποία έχει ε, λιγότερε επιπτώσει από τον άνθρακα. θεωρούμε ότι είναι κοινέ οι θέσει που έχουμε εδώ στο πάνελ και θεωρούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει και διάλογο με τι ενδιαφερόμενε χώρε, διότι ο καλό διάλογο αποτελεί και το σημείο κίνηση για να ξεκινήσουμε. Ε, Σα ευχαριστώ και πάλι. Ήταν πολύ επικοδημητικά τα όσα ακούσαμε από πλευρά Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ. Να δώσουμε τώρα το λόγο στου εμπειρογνώμονε για να απαντήσουν στι παρατηρήσει των Ευρωβουλευτών και τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πριν δώσω το λόγο στον κύριο Νόιζερ για να ολοκληρώσει. Πέντε λεπτά για την απάντησή σας. Ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Όσον αφορά την περίπτωση της Ταϊλάνδης, δεν κοιτάξαμε συγκεκριμένα την χώρα αυτή. Κοιτάζαμε στην έρευνα την υποσαχάρια Αφρική και την Ινδία. Αυτό που βγήκε από την έρευνα είναι ότι οι χώρες που έχουν την ε, μεγαλύτερη πρόοδο έχουν μεγαλύτερη εθνική προτεραιότητα στην πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια πρωτίστω και ενέργεια γενικότερα και ο στόχο είναι να υπολογίσουμε το κόστο. Και φυσικά αυτό που επακολουθεί είναι οι σχετικέ μακροοικονομικέ και δημοσιονομικέ πολιτικέ και αναφέρθηκε ήδη πριν το τοπικό κίνητρο για να αποδεκτούν τις ε, τεχνολογίες αυτές και να τις κρατήσουν μακροπρόθεσμα βιώσιμες. Όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση, Ισχύει ότι η ενεργειακή απόδοση μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στην αύξηση πρόσβασης ε, στην ενέργεια. Θα έλεγα όμως ότι όσον αφορά τα έργα που υπάρχουν τώρα, το φράγμα Κοσόμπο στην Κάνα, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Παγκόσμια Τράπεζα και αύξησε την απόδοση, την ενεργειακή απόδοση κατά 31%. Βλέπετε δηλαδή τη διαφορά. Αυτά τα έργα μεγάλης κλίμακας δεν έχουν τόσο μεγάλο αντίκτυπο στις ε, κοινωνίες της υπαίθρου. Η ενεργειακή απόδοση δεν είναι λοιπόν φλέγον θέμα προς το παρόν. Το θέμα είναι να υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια. Δεν θα εστίαζα λοιπόν τόσο πολύ στην ενεργειακή απόδοση κατά από αυτό το πλαίσιο όχι λοιπόν τόσο σημαντική στα ε, έργα μικρής κλίμακας στην Ήπεθρο. Ε, εκεί λοιπόν ε, είναι ο στόχος μας σε αυτή την έρευνα. Δεν ξέρω αν η συναδελφός μου θα ήθελε να προσθέσει κάτι. Ναι, το πρόγραμμα Energy Stop είναι ένα πρόγραμμα στις Ηνωμένε Πολιτείε. Υπάρχει όμως συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο προϊόντων διαθέσιμα και στις Ηνωμένε Πολιτείε και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό που ήθελα όμως ε, να πω δεν είναι ότι είναι μάλλον ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα πρέπει να επιδείξουν σοφία όσον αφορά την ε, ενεργειακή απόδοση στις χώρες τους. Διαφορετικά κινδυνεύουν να μην λάβουν τα προνόμια τα οποία θα μπορούσαν να λάβουν. Και επίσης εταιρείε, για παράδειγμα, που παράγουν μονάδες κλιματισμού, ενδεχομένως να ξεφορτωθούν τα προϊόντα που σπαταλούν μεγάλη ενέργεια στις ε, χώρες αυτές αντί να τα πουλήσουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική. Δεν Μίλησα λοιπόν πιο πολύ από πλευράς ε, προσφοράς. Αυτό ήθελα να πω με, με τη χρήση προϊόντων ενεργειακής απόδοσης. Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ και εγώ τους εμπειρογνώμονές μας. Πιστεύω πως σε γενικές γραμμές συμφωνείτε με την έκθεση και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα σχόλιά σας. Θα προσπαθήσω να τα ε, υιοθετήσω και να τα λάβω υπόψη. Πράγματι, η ενεργειακή απόδοση είναι σημαντική. Χρειαζόμαστε πρόσβαση σε ενέργεια καθαρή, αξιόπιστη, βιώσιμη και αποκεντρωμένη και επίσης προσιτή οικονομικά. Εμείς μπορούμε να, ε, να δώσουμε την ενέργεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Το θέμα είναι αν οι άνθρωποι αυτοί θα μπορούν να την πληρώσουν. Αυτό είναι το θέμα. Οι κυβερνήσεις με τις οποίες ε, έχουμε συζητήσεις χρειάζονται ε, ισχυρές... Χρειάζεται ισχυρή διαπραγματευτική θέση. Η σημασία του ιδιωτικού τομέα, όπως αναφέρθηκε και από την Κομισιόν, είναι μεγάλη. Αναφέρθηκε ότι από 20 πρέπει να γίνει 80% συμμετοχή σε ιδιωτικών φορέων. Οι ιδιωτικοί φορείς λοιπόν πρέπει να αναμειχθούν και αυτοί στην ε, παροχή ενέργειας. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι η πρόσβαση στην ενέργεια αποτελεί την σύνδεση στους, ε, με τους στόχους της ε, χιλιετίας. Τους στόχους από το 2015 και μετά Συνολικά χρειαζόμαστε να καταβάλουμε μεγάλες προσπάθειες και αυτό το κατέστησαν σαφές οι εμπειρογνωμονές μας. Χρειαζόμαστε να καταβάλουμε πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ. Merci beaucoup. Ευχαριστούμε, λέει πρόεδρε. Σα θυμίζω ότι η προθεσμή για τις τροπολογίες πρόκειται να εκπνεύσει στις 16 Ενδεκάτου το μεσημέρι. 16 11 το μεσημέρι. Και 8 Δεκεμβρίου θα γίνει η ψηφοφορία. Και τώρα περνάμε στο σημείο παραγμό 15 της Μεσής Διατάξεως. Πρώτη για την ε, έκθεση ε, Birgit Schnieber Γιάστραμ. Το θέμα είναι η σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι αναδυόμενες χώρες. Βραζιλία συγκεκριμένα, Ρωσία, ε, Νότιος Αφρική και Ινδία. Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Νότια Αφρικανική Ένωση, επομένως δεν είναι θέμα βέβαια καθαρά ανάπτυξης, όμως είναι θέμα γενικότερο και αφορά τη θέση μας, τις σχέσεις μας όσον αφορά την εξωτερική πολιτική, οπότε ευθύς αμέσως θα δώσουμε την ε, ε, σκητάλη στην κυρία Σνίμπερ Γιάστον, ούτως ώστε να μας παρουσιάσει την έκθεση και επίσης πρέπει να ευχαριστήσουμε και τους ε, εμπειρογνώμονες, τους ειδικούς, τα θέματα συνέργειας οι οποίοι τώρα την αίθουσα. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η σχέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης με, τα, με τις χώρες BRIC πιστεύω πως έχει μια ιδιαίτερη σημασία. Αν δούμε ένα ερωτηματολόγιο που έγινε στη Γερμανία. Σύμφωνα με αυτό, 97% πιστεύουν ότι η Κίνα έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην αγορά. 91% των ερωτηθέντων αποκαλούν την Κίνα μεγάλο επενδυτή. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για μας 76% θεωρούν την Κίνα εταίρο που θα βοηθήσει στη λύση των παγκόσμιων προβλημάτων και αυτό δεν φαίνεται μόνο και από την ε, σύναψη στρατηγικών συνεργασιών. Οι χώρες BRIC δεν είναι ένα συμπαγές μπλοκ αλλά είναι ένα δίκτυο. το οποίο αποφασίζει από κοινού για κάποια πολύ σημαντικά ζητήματα και οι συνέπειε για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κοινή πολιτική. Πρέπει να βρούμε κοινά σημεία για μια πολιτική απέναντι σε αυτές τις χώρες. Το θέμα είναι, ότι, το, θέμα είναι το εξής. Πού θα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας. Στην Κίνα, για παράδειγμα. Ξεκάθαρο είναι ότι ορισμένες χώρες BRIC προτιμούν αυτή την τακτική που ακολουθούν από ότι μια παγκόσμια κοινή στάση. Τι θέλουμε εμείς να κάνουμε, θέλουμε να εμβαθύνουμε τη συνεργασία. Θέλουμε να κρατήσουμε τις αξίες μας, θέλουμε να διευρύνουμε τις αξίες μας. Αν θέλουμε να διευρύνουμε τις αξίες μας πρέπει να εργαστούμε γι' αυτό. Στην... Όσον αφορά τη συνεργασία υπάρχουν πολλά που υπολείπονται. Για παράδειγμα, ο γόνα κατά του AIDS, ο, ε, διάλογος διάλογο όσον αφορά τον προπολογισμό, η συνεργασία για τα ερευνητικά προγράμματα. Μία παραπάνω δυνατότητα για την εμβάθυνση της συνεργασίας ή τουλάχιστον για μια συντονισμένη συνεργασία θα μπορούσε να έχει ως κόνσεπτ την ε, ανάπτυξη την αποδοτική ανάπτυξη. Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, εξαιτία τη θα μπορούσα να αναλύσω αυτά τα σημεία στις ε, τροπολογίες. Για παράδειγμα, τον τριμερή διάλογο, την ε, συνεργασία για καλύτερη, καλύτερη μακροοικονομική συνεργασία την εταιρική κοινωνική ευθύνη. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα που δεν είναι απαραίτητα πολιτικά. Χρειάζονται πολύ περισσότερες έρευνες και εκθέσεις εμπειρογνωμόνων. Σε επίπεδο κρατών μελών φυσικά είναι πολύ σημαντικό. Είμαι ευγνώμων για τις ε, προτάσεις που έχετε, που ενδεχομένω έχετε. Η αλλαγή της παγκόσμιας τάξης τώρα με, την, ε, με, τα, τις χώρες BRIC θα μπορούσε να είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για μας, αλλά πρέπει να αποφασίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία αυτή που μας δίδεται. Merci beaucoup. La parole est à Madame Keller. Ευχαριστούμε Κέλλερ. Ευχαριστώ πολύ. και Ευχαριστώ πολύ για την έκθεση. Πιστεύω πως είναι μια πάρα πολύ καλή αρχή για τις τροπολογίες που θα κληθούμε να κάνουμε για να ξεφορτωθούμε αυτή την... αυτό τον περιορισμό της μιας σελίδας. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ σε ορισμένα ζητήματα τα οποία πιστεύω πως ακόμα λείπουν ή δεν αναλύονται όσο θα έπρεπε στην έκθεση. Περιοχές που νομίζω ότι η συνεργασία είναι, πολύ, είναι αναγκαία στην κλιματική αλλαγή, στην μεταφορά τεχνολογίας, στην βιώσιμη ανάπτυξη, στην ε, διαδικασία ριοσύν. θα πρέπει να δούμε πώς θα διασφαλίσουμε κοινωνικά στάνταρ και περιβαλλοντικά στάνταρ επίσης. Γνωρίζω ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες δεν χαίρονται πολύ με την προοπτική του να βάλουν αυτά, αυτά τα, να λάβουν αυτά τα πράγματα υπόψη. Αυτό όμως που θα μπορούσαμε να δούμε στη συνεργασία μας με τις χώρες BRICS είναι η καλύτερη, ο καλύτερος συντονισμός της παγκόμιας διακυβέρνησης, να χρησιμοποιήσουμε πολυμερή φόρουμ αντί για διμερή φόρουμ, Επίσης, πιστεύω πως οι χώρες BRIC θα είναι ζωτική σημασία στην μεταρρύθμιση της οικονομικής διακυβέρνησης και αυτό είναι ένας τομέας που νομίζουμε ότι εσείς μαζί με τις χώρες BRIC θα, μπορέσετε να, θα μπορούσατε να επεξεργαστείτε περισσότερο. Πιστεύω πως τώρα με, τις, ε, με το φόρουμ υψηλού επίπεδου είναι μια καλή ευκαιρία να χρησιμοποιήσουμε αυτό το φόρουμ για καλύτερη συνεργασία με τις χώρες BRIC, γιατί ξέρουμε ότι υπάρχουν ακόμα δυσκολίες και ότι πολλές χώρες αυτές διστάζουν. Θα πρέπει λοιπόν να προσπαθήσουμε να κάνουμε τις χώρες BRIC να συμφωνήσουν μαζί μας, να έρθουν με το μέρος μας, αλλά και να τους δώσουμε κάτι σε αντάλλαγμα, μεγαλύτερο βάρος στους παγκόσμιους οργανισμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μπέρμαν έχει το λόγο. Θα είμαι πολύ σύντομος, διότι ο σκιώδης εισηγητής, ο κύριος Κάσμαν, δεν είναι εδώ σήμερα και θα ήθελα να πω ότι ακούγοντας ε, την έκθεση αυτή, θεωρώ ότι συμφωνούμε στο 99% των θεμάτων. Αυτό μόνο. Το μόνο το οποίο θα ήθελα να προσθέσω σε προσωπικό επίπεδο είναι ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να φοβόμαστε αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες. Οι χώρες αυτές ε, θέλουν να γίνουν μεγάλες οικονομικές δυνάμεις και ε, αναμφίβολα να γίνουν και ανταγωνιστές μας. Ναι, αλλά θα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα και πελάτες. Και σε θέματα αναπτυξιακής βοήθειας θα πρέπει να τους βλέπουμε ως εταίρους και όχι αντιπάλους που θέλουν να εφαρμόσουν ένα διαφορετικό πρόγραμμα. Ε, έχουμε όλοι να κερδίσουμε αν έχουμε με ε, εταίρους όπως την Κίνα και την Ινδία. Η Βραζιλία, για παράδειγμα, έχει ένα τελείως διαφορετικό ανεπτυξιακό πρόγραμμα με τη Ρωσία. Ε, ο Μετβέργεχ και ο Πούτιν έχουν τελείως διαφορετικά προγράμματα και διαφορετικούς στόχους και ε, διαφέρει και το πρόγραμμά του από το πρόγραμμα τη Νοτιού Αφρική. Δεν μπορούμε να τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι απλώ και μόνο διότι πρόκειται για πέντε οικονομίε, οι οποίε αυξάνονται και αναπτύσσονται συνεχώ ε, και μόνο αυξάνονται. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να λάβει το λόγο. Oui. Καλησπέρα σας. Να συστηθώ. Ανδρέα Μόνη. Είμαι συντονιστής πολιτικής για το Τμήμα Παγκοσμίων Θεμάτων της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης. Καταρχάς, να σας πω ότι χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να ετοιμάσει μια έκθεση για το θέμα αυτό, το οποίο είναι στρατηγική σημασία για μας Επίσης, χαιρετίζω το γεγονός ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σωστά ενετόπισε κατά την άποψή μου τα πιο σημαντικά στοιχεία αυτής της συζήτησης και τονίζει τις πιο σημαντικές αρχές οι οποίες θα πρέπει να διέπουν ε, τη σχέση μας ε, με τις χώρες ε, BRICS ιδίως την έννοια της πιο ελαστικής προσέγγισης όπως ανέφερε και ο προλαλής σας, πρέπει να διαφοροποιήσουμε την προσέγγιση μας, πρέπει να είμαστε ευέλικτοι και επίσης θα πρέπει να έχουμε και μια ολοκληρωμένη προσέγγιση η οποία θα λαμβάνει υπόψη και το γεγονός ότι είναι πολύ περίπλοκες οι πραγματικότητες της κάθε μίας από αυτές τις αναδυόμενες οικονομίες και σε κάποιο βαθμό ακόμα είναι αφενός αναπτυσσόμενες χώρες αλλά αφετέρου ε, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με πολύ δυναμικές ε, οικονομίες και με πολύ σημαντικές ε, τεχνολογικές, ε, πολιτιστικές και ρυθμιστικές πραγματικότητες. Επομένως, η διαφοροποιημένη προσέγγιση από πλευράς μας είναι ουσιώδης και η τρίτη βασική αρχή που θα πρέπει να διέπει τις σχέσεις μας είναι ότι θα πρέπει να βλέπουμε και στο μέλλον για μας ε, να έχουμε, το να έχουμε σχέση με τις BRICS ε, σημαίνει ότι επενδύουμε και στο μέλλον. Όπως ανέφερε και ο προλαλής σας λοιπόν ότι θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι δημιουργούνται νέες πραγματικότητες οι οποίες ε, είναι ήδη πολύ σημαντικές διότι οι χώρες αυτές είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες στο διεθνές προσκήνιο και είναι πολύ αποτελεσματικοί παράγοντες σε πολυμερή και παγκόσμια ζητήματα. Αναφέρομαι για παράδειγμα στο ρόλο τους ε, στα Ηνωμένα Έθνη, το ρόλο τους στο G20 όπως ε, τον διαπιστώσαμε προσφάτως, το ρόλο τους ε, στη νότια-νότια συνεργασία και επίσης σε περιφερειακές οργανώσεις τις οποίες ανήκουν. Θα πρέπει λοιπόν να επενδύσουμε στις χώρες αυτές ως εταίρους μας θα πρέπει να συνομιλούμε μαζί τους, θα πρέπει να ε, κάνουμε σύγκριση των αξιών μας με τις αξίες τους οι οποίες διαφέρουν, αλλά θα πρέπει να ε, παρέχουμε και εμείς κάποια στοιχεία σε αυτή τη συζήτηση, ένα επιπρόσθετο όφελος, ε, μια δική μας συνεισφορά. Υπάρχει βεβαίως ένα μοντέλο το οποίο θα μπορούσε να ε, τους ενδιαφέρει, μπορούν να μας μιμηθούν, υπάρχει ένα ρυθμιστικό πλαίσιο, το κοινοτικό κεκτημένο, το οποίο θα μπορούσε ίσως να τους ενδιαφέρει. Επιπλέον, θα πρέπει ε, να ε, τους πείσουμε να συμμετέχουν σε παγκόσμια θέματα. Ε, πολύ σωστά αναφέρθηκε προηγουμένως η κλιματική αλλαγή, το περιβάλλον βεβαίως, οι μεταφορές, η ενεργειακή απόδοση, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία ενδιαφέρουν ιδιαίτερα το G20. Ολοκληρώνοντας να σας πω ότι ο Διευθύνων Συμβουλός μου, ο κύριος Λέφλερ, θα παρουσιάσει την επίσημη θέση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις χώρες αυτές στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Κοινοβουλίου και ε, είναι ο καθήλυν αρμόδιος για να σας παρουσιάσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Η Ευχαριστώ θερμά τους συναδέλφους για τα σχόλιά τους ε, και για την παρατήρηση της κυρίας Κέλλερ. Συμφωνώ για την διατηρήση των ευρωπαϊκών αξιών. Πρέπει να δούμε όμως και τις ε, άλλες κουλτούρες και να δούμε ε, εάν μήπως εμείς είμαστε κάπως αλαζόνες, εάν θεωρούμε δηλαδή αυτούς καλύτερους. Πρέπει να δούμε λοιπόν εάν η κριτική αυτή τη στιγμή είναι αναγκαία ή όχι και εάν ίσως θα έπρεπε καλύτερα να επικεντρωθούμε σε προς, τις προσπάθειες ε, στις αναπτυσσόμενες εκείνες χώρες οι οποίες δεν έχουν το δικό μας επίπεδο. Πρέπει να δούμε ότι αυτές οι συζητήσεις είναι καλό να γίνουν επίσης όρις και να γίνουν σεβαστές οι διαφορετικές απόψεις. Και εκεί βρίσκονται οι ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ, λέει η Πρόεδρος, και σας υπενθυμίζω ότι η προθεσμία κατάθεση των ε, τροπολογιών εκπνέει στις 10 Νοεμβρίου το μεσημέρι και η, ψήφιση θα γίνει στις 5-12 του. Και τώρα πάμε στο σημείο 16 της σημερινή διατάξεως. Είναι η έκθεση τη Ιζαμπέλα Λέβιν και αφορά την Αλληλευτική Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Γουινέας Μπισάου. Η σκητάλη στην ε, μεγάλη μας εμπειρογνώμονα, την Ιζαβέλα Λόβεν, για τα θέματα αλληλείας. Ε, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ναι, θα μιλήσουμε για άλλη μία από τις διάφορες αλήθειες συμφωνίες που έχουμε με αναπτυσσόμενες χώρες, ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ουενέμπισό είναι μία από τις λιγότερα αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Ε, τα δύο τρίτα των οικοκυριών είναι κάτω από το ορίο της φτώχειας. Και επίσης ε, παρά την αναπτυσσόμενη χώρα και έχει πρόβλημα, δεν πλήττει τα κριτήρια για τις ενισχύσει τη Παγκοσμίας τράπεζα. Και η Αλία εξελίσσεται αυτό του όμως παρόλα αυτά, ακριβώς όσον αφορά τις ψηλούς πόρους, είναι μια πλούσια χώρα. Είναι δύο φορές πιο μεγάλη η θαλάσσια επικράτηση τη από την, το, το έδαφος, την εδαφική. Να λοιπόν, ποια είναι η πηγή όλων αυτών των ε, αλληλευτικών πόρων. Έχουν μικρά πελαγικά, έχουν μεγάλα μεταναστευτικά, ε, κεφαλόποδα, τόνο, γαρίδες και, και, και μιλούμε για 12.000 αλληλείς οι οποίοι εκεί πέρα ε, είναι παραδοσιακή αλληλείας και ε, αλλιεύουν και όχι αυτούς που κάνουν παράπλευρα δραστηριότητα, δεν τους υπολογίζουμε. Επειδή δεν έχουν άλλου είδου ε, τροφή για, για πρωτενη, καταλαβαίνουν πάρα πολύ ε, ε προϊόντα. Οπότε έχουμε εδώ πέρα αυτή τη συμφωνία και στις 15 Ιουνίου 2010 έληξε αυτή η προηγουμένη συμφωνία και έχουμε τώρα ένα νέο πρωτόκολλο το οποίο καλύπτει μια περίοδο ενό έτου. Από το 16 Ιουνίου 2011 και από τότε ισχύει σε προσωρινή βάση. Οπότε έχουμε αυτό το νέο πρωτοκόλλο το οποίο δεν τροποποιεί τις ε, δυνατότητες για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επίσης ε, έχει την διαπρικοδότηση όπως το προηγούμενο. 7.500, 7.500.000 για αυτό το έτος. Και αυτό αντιστοιχεί στις αδειοδοτήσεις 37 αλληλευτικών τόνου και επίσης και σε άλλες στρώτες. Και μιλάμε για 8.800 τόνους μεικτού τονάζ για αυτά τα σκάφη. Επομένως έχουμε 4,5 εκατομμύρια ε, ευρώ που με αυτά αγοράζουν δυνατότητα προσβασιμότητας και επίσης έχουμε 2,5 εκατομμύρια περίπου τα οποία αφορούν ένα άλλο επιπλέον κονδύλι το οποίο αφορά την αναπτυξιακή ενίσχυση για, την, ε, ε, για τον στην χώρα. Μισό εκατομμύριο ευρώ επίσης ε, αφορούν την θέσπιση ενός συστήματος υγείας και φυτογενομικής κάλυψης για τα προϊόντα της αλίας. 35% λοιπόν από αυτήν όλη την χρηματοοικονομική συμβολή την προβλέπουμε ούτως ώστε να καλυφθεί ο αληθικός τομέας στη χώρα. Έχει γίνει μια μελέτη αξιολόγηση όσον αφορά αυτήν την ελευθερική συμφωνία και προέκυψε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μάλλον ε, σε περιορισμένο βαθμό αλλά έχει θετική σχέση σχέση αποτελέσματος η ενίσχυση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια για τη χώρα Μιλάμε για 7,3% του συνόλου του προπολογισμού του κράτους. Και μιλούμε για 88% της δαπάνης επί τη βάση του προπολογισμού για την αλία. Άρα, για την οικονομική σταθερότητα τη χώρα είναι κάτι το πάρα πολύ σημαντικό αυτή η ενίσχυση. Αυτή η αξιολόγηση επίση κατέληξε σε κάποια άλλα ζητήματα. κάποιες διατάξει που δεν είχαν εφαρμοστεί με τον καλύτερο τρόπο. Φερρυπίν έχουμε πάρα πολλές απορρίψεις. Κυρίως όσον αφορά τη γαρίδα. Ούτε συμμορφώθηκαν τα γενικά σκάφη με τις υποχρεώσεις ε, ειδοποίησει όταν βγαίνουν από τα χωρικά έδρα της χώρας σε σχέση με το τι αλλήλων έχουν. Και όλα αυτά επιδέχονται βελτίωση. Έχουμε τώρα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξη και έχουμε και κάποια εκ των υστέρων αξιολόγηση που κατέληξαν ότι οι αρχές της χώρας και η Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν και συνεχίζουν πολιτικό διάλογο και συνεργάζονται όσον αφορά τη βελτίωση της ελληνικής πολιτικής. Που επιδέχεται βελτίωση. Πάντω είπαμε ότι η μακροοικονομική σταθερότητα τη χώρα στηρίζεται πάρα πολύ αυτή την ενίσχυση και σε αυτό το νέο πρωτόκολλο έχουμε κάποιε νέε διατάξει όσον αφορά τι καταβολέ αυτή τη οικονομική ενίσχυση που εάν έχουν παραβίαση των δικαιωμάτων θα ανασταλεί. Επίσης θα υπάρχει αναστολή εάν η γωνία Μπισάου δεν μπορέσει να αποκτήσει βιώσιμη ελεία. Και αυτό πάρα πολύ θετικό. Και σε σχέση με το μέλλον αυτή τη συμφωνίας θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και η Ευρωπαϊκή Ένωση στα σοβαρά να το δουν, να παρακολουθήσουν το τι γίνεται με την εφαρμογή της συμφωνίας. Να γίνουν πράγματα όπως προβλέπει το πρωτόκολλο. Και μια βασική αρχή είναι ότι τα σκάφη της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πηγαίνουν μόνο εκεί που υπάρχουν πλεονάσματα, εκεί που δεν ε, ψαρεύουν οι ντόπιοι, εκεί που δεν χρειάζεται οι ντόπιοι να ψαρεύσουν για να τραφούν. Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τέτοιες ε, διαδικασίες ώστε να αποκλείεται η λαθραλίευση να υπάρχει διαφάνεια μια που, μια που έχουν τόση θάλασσα επικρατεία εκεί που είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει έλεγχος. άλλο. Θα πρέπει αυτό να αντιμετωπιστεί άμεσα. Είναι μεγάλες προσέντες παραλίευματος και των όπως είπαμε, όσον αφορά των απορρίψεων όσον αφορά τις, ε, τις γαρίδες. Εκεί μπορούμε να πάμε στο 85% του συνόλου του ελεύματος που ξαναπετάνε μέσα στη θάλασσα. Όλα αυτά είναι, είναι πρωτεΐνη, πολύτιμη που θα μπορούσε κανείς να την πουλήσει τοπικά και τώρα με κάποιο είδου περίεργη, λογική των, των σκαφών της Ένωσης απορρίπτουν τη θάλασσες. Υπάρχει επίση κάποια κοινή επιτροπή που προβλέπει αυτό το πρωτόκολλο, σύμφωνα με το οποίο η Ένωση και η Γουινέα Μπισάου πρέπει να φροντίσουν την ορθή εφαρμογή του πρωτοκόλου. Και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα τη διαφθοράς. Και τα χρήματα πηγαίνουν εκεί που πρέπει. Άλλο πρόβλημα που έχει σχέση με αυτή την αξιολόγηση είναι ότι κάποια γενοτικά σκάφη αλλιεύουν με άλλη σημαία. Αλλάζουν τη σημαία και έτσι αποφεύγουν κάποιες υποχρεώσεις. Δεν θα πρέπει να τους επιτρέπεται ε, να ξαναγυρίσουν στα κοινωτικά νεολόγια. Και έτσι να διατηρηθεί η ρήτρα αποκλειστικότητας. αυτό το γράμμα και το πνεύμα του νόμου να τηρείται. Τέλος. Θα πρέπει να γίνεται μια αιτήσια έκθεση και να υποβάλλεται στο Κοινοβούλιο σε σχέση με το πώς πάει, πώς εφαρμόζεται αυτό το πρωτοκόλλο και έτσι να έχουμε διαφάνεια. Και πιστεύω όπως και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Πρόσωπη της Αλίας ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί αυτή η σχέση μεταξύ Γουνίας Μπισάου και Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι να βελτιωθεί η αλληλευτική πολιτική στη χώρα και να καταπολεμηθεί η λαθραλήψη που είναι πολύ σημαντικό πρόβλημα. Αν επομένως εφαρμοστεί ορθά αυτό το πρωτόκολλο, θεωρώ ότι είναι σωστό το να δοθεί η παράταση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ διότι επιμείνατε και στη σημασία των ελέγχων και θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η Γουινέα Μπισάου διαθέτει λιμενικές αρχές ε, για να μπορούν να ελέγχουν επί τόπου τα πράγματα. No. Uh, Η κυρία Λεβίν, όχι. Υπάρχει το κέντρο ελέγχου στο Βίγκο, το οποίο συντονίζει τις υπηρεσίες ελέγχου των κρατών μελών, ώστε να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους πόρους τους καλύτερα, αλλά δεν υπάρχουν ίδια σκάφη, τουλάχιστον προς το παρόν. Μπορούν να αναβλώσουν ένα σκάφος ε, το οποίο ελέγχει λίγο τον Ατλαντικό στην πράξη αλλά δεν πηγαίνει μέχρι κάτω στη Δυτική Αφρική. Ίσως λοιπόν θα μπορούσε να επενδύσει σε κάτι τέτοιο η Ευρωπαϊκή Ένωση για να προσπαθήσει να δώσει απτή βοήθεια για την ε, ε, φύλαξη αυτών των ε, λιμένων, διότι πραγματικά η λαθραλίευση αποτελεί μάστιγα. Ευχαριστώ ρόγο στον, επίτροπο, στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Πέρκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και την εισηγήτρια για την πληρέστατη παρουσίασή της για το πρωτόκολλο αλληλευτικής συμφωνίας με τη βουινεα Μπισάο. Νομίζω ότι τα βασικά ακούστηκαν. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συμφωνία και για το στόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, διότι υπάρχουν πολλά αλληλευτικά είδη που μας ενδιαφέρουν, πολλά σκάφη συμμετέχουν, πολλές χώρες μέλη συμμετέχουν, αλλά πρόκειται και για μια συμφωνία η οποία είναι ζωτική σημασία για τη χώρα, δηλαδή για τη βουινεα Πισάο, η οποία έχει πολύ σημαντικούς ε, πόρους ε, που εξαρτώνται από την αλληλευτική συμφωνία και για τη σταθερότητα της χώρας, αλλά και εξαιρετικά ε, σημαντικό για τη συμφωνία της υπηρεσίας του Υπουργείου Αλληλείας και για τους πόρους που διατίθενται σε θέματα διαχείρισης και εποπτείας της αλληλείας. Ήθελα εδώ να σταθώ αμέσως στην ερώτηση που διατυπώσατε για τις μονάδες επιφυλακής. Με τη Γουινέα Μπισάου ε, υπάρχουν κάποια σκάφη τα οποία μόλις αγοράστηκαν από το Υπουργείο. Κάποια ήδη ε, χρησιμοποιούνται. Ε, έχουν χρηματοδοτηθεί βάσει του Ταμείου και άλλα ε, σκάφη τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για την λιμενοφυλακή των ακτών της Γουινέα Μπισάου. Πρόκειται για μικρά σκάφη τα οποία θα συνεισφέρουν τουλάχιστον για την ε, ε, περιφρούρηση του αρχιπελάγους ε, και των λιμένων. Υπάρχουν επίσης στρατιωτικές δυνάμεις οι οποίες είναι διαθέσιμες στη Γουινέα Μπισάου για μεγαλύτερη περιφρούρηση αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ρόλος του στρατού αμφισβητήθηκε τα τελευταία χρόνια ε, διότι θέλουμε να ε, υπάρχουν αντικειμενικές αυτόνομες μονάδες περιφρούρησης που θα ανήκουν στη Υπουργείο Αλληλείας ώστε να μην υπάρχει εξάρτηση από το στρατό. Θα ήθελα να επαλέλθω εν συντομία και στο θέμα των ε, πόρων. Να σας πω ότι ο στόχος στη συμφωνία αυτή είναι να αλλιεύεται μόνο το πλεόνασμα, δηλαδή ό,τι δεν αλλιεύεται από τους ε, αλληλείς τοπικά και δεν ε, θέλουμε φυσικά να υπάρχει κανένας αντιγωνισμός μεταξύ του ερασιτεχνικού αυτού στόλου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, και του ευρωπαϊκού στόλου, ο οποίος ε, ούτως ή άλλως αλλιεύει αρκετά μεγάλο απόθεμα και αλλιεύουν και σε πιο απομακρυσμένα ύδατα ε, σε σχέση με τα ύδατα κοντά στις ακτές τα οποία αλλιεύουν οι παραδοσιακοί αλλοίς. Όσον αφορά τις κατηγορίες που αναφέρθηκαν, δηλαδή ε, τα κεφαλόποδα και τις γαρίδες, ε, δεν χρησιμοποιούνται όλα τα ποσοστά που έχουμε ε, από, τις, από τον Ευρωπαϊκό Στόλο. Χρησιμοποιείται ένα 45%, επομένως μένει ένας πολύ μεγάλος αριθμός όσον αφορά τώρα τα αθηνοειδή που προβλέπονται στη συμφωνία αυτή και εκεί είναι πολύ μικρότερος ακόμα ο κίνδυνος ανταγωνισμού διότι η ε, Γουινέα Μπισάου δεν έχει θυναλιευτικά, επομένως δεν μπορεί να αλλιεύσει τόνους. Εμάς μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα η παρακολούθηση της συμφωνίας και η συνέχεια. Πρόκειται για μια συμφωνία την οποία έχουμε παρακολουθήσει περισσότερο από όλε ίσω. Ε, υπάρχει και η μεικτή Επιτροπή η οποία προβλέπεται να συνεδριάσει την επόμενη εβδομάδα στις Βρυξέλλες και ε, θα έχουμε σε σύνολο τρεις ε, μεικτέ επιτροπέ εντό του 2011 για τη συνέχεια αυτή τη συμφωνία. Ε, αυτό νομίζω ότι αποδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η συμφωνία και σε πολυτεμιακό επίπεδο, διότι γνωρίζουμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν αρκετέ καθυστερήσει, υπήρξαν αρκετέ δυσκολίε οι οποίε ε, είχαν σχέση και με τι πολιτικέ αλλαγέ, ε, τι δυσκολίε τη κυβέρνηση τη Γουινέα Μπιχάου να απορροφήσει τα κονδύλια. Αλλά στόχος μας είναι να τους υποστηρίξουμε κατά τρόπον ώστε να μπορούν να δαπανηθούν αυτά τα κονδύλια με αποτελεσματικό τρόπο και θα μπορούσαν να δοθούν και κάποια παραδείγματα για το τι έχουμε κάνει. Υπάρχει σύστημα VMS, το δορυφορικό σύστημα παρακολούθησης των σκαφών και ε, υπάρχουν και αρκετά ε, θέματα εποπτείας ε, βάσει των σκαφών αυτών και νομίζω ότι το α είναι να υπάρχει ακριβώς το VMS επί των σκαφών για να εποπτεύουμε τι γίνεται. Στη Γουινέα Μπισάο πριν από κάποιες εβδομάδες ε, μπόρεσαν να δω η διεισόμαση τι ακριβώς γίνεται στους λιμένες. Ε, Υπάρχει ένας ε, λιμένας ο οποίος δεν χρησιμοποιείται σχεδόν καθόλου από τις αρχές της Γουινέα Μπισάου και επομένως θα μπορούν ίσως να εκφορτώνουν εκεί τα θυναλιευτικά. Υπάρχουν προκυμές, υπάρχουν και κατάλληλες υποδομές οι οποίες χρησιμοποιούνται και για μεταποίηση και έχει ολοκληρωθεί πλέον η κατασκευή του νέου λιμένα και θα είναι στη διάθεση των ευρωπαϊκών σκαφών. Τώρα, η διαφορά που είχαμε σε πολιτικό επίπεδο ε, σε σχέση με την προηγούμενη συμφωνία είναι ότι καταφέραμε να εντάξουμε και μία ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό ε, ουσιαστικά επιτηρούμε επί της χώρας και ελέγχουμε πώς έχει κατάσταση και αν η κατάσταση σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, και δημοκρατίας ε, επιδεινωθεί θα μπορέσουμε να αναστείλουμε την εφαρμογή του πρωτοκόλου. Ε, νομίζω ότι δεν υπάρχει βέβαια πρόβλημα διότι αντίθετα με τις προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου αναφέρομαι στην απόφαση του Συμβουλίου της 18 Ιουλίου φαίνεται ότι υπάρχει πολύ σημαντικό ε, ποσοστό προόδου σε θέματα διακυβέρνησης. Αυτό το επιβεβαιώνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι διαβουλεύσεις που έγιναν για το άρθρο 96 νομίζω ότι μπορούν να ολοκληρωθούν. Υπάρχει μια ρήτρα παρακολούθησης η οποία συνεχίζει να είναι ενισχύ βεβαίως αλλά ε, νομίζω ότι έχουμε γυρίσει σελίδα και μπορούμε πλέον να έχουμε πολύ πιο σημαντικές ε, σχέσεις, πολύ πιο υγιείς σχέσεις με την Γουινέα Μπισάου και σε θέματα ε, διαχείρισης της αλληλείας, τα όσα είχαμε στην αλληλεία τα τελευταία χρόνια, ε, ο υπεύθυνο, ο Υπουργός ε, φεύγει από τη θέση του και θα τον αντικαταστούσει μια νέα πολιτική προσωπικότητα στη Γουινέα Μπισάου. Δεν θα ήθελα να μονοπολίσω το χρόνο της ε, συνεδρίασής σας. Ε, η ρήτρα που αναφέρατε και εσείς είναι πολύ σημαντική. Τα ευρωπαϊκά σκάφη θα πρέπει να λιεύουν μόνο βάσει αυτής της συμφωνίας, έτσι ώστε να υπάρχει ε, κατάλληλος έλεγχος και διαφάνεια. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Αυτές ήταν οι παρατηρήσεις μου, οι οποίες ελπίζω να συνεισέφεραν και στη συζήτηση. Ευχαριστώ. Η κυρία Λεβίν για να ολοκληρώσει. Uh, yes. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση και για τις επεξηγήσεις σας. Χαίρομαι πολύ που μαθαίνω ότι η Γουινέα Μπισάου τώρα έχει αγοράσει σκάφη ελέγχου. Γιατί όταν επισκέφτηκα τη χώρα αυτή πριν από λίγα χρόνια είχαν μόνο δύο σκάφη και το ένα δεν λειτουργούσε καν. Δεν μπορούσαν να πληρώσουν και τα καύσιμα βασικά. Και ήταν λοιπόν στο λιμάνι. Συμφωνώ λοιπόν ότι ε, το OVMS είναι μια σημαντική βελτίωση και ότι χωρίς αυτό δεν γίνεται να διεξαχθεί κανένας έλεγχος. Και επίσης χάρηκα πολύ που άκουσα ότι συμμορφώθηκε η χώρα με την ε, ερήτρα της αποκλειστικότητας. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για τις πληροφορίες σας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Να σα υπενθυμίσω ότι η προθεσμία κατάθεσης τροπολογιών είναι η 10η Νοεμβρίου στι 5 το απόγευμα και η ψηφοφορία θα γίνει στι 8 Δεκεμβρίου. Η επόμενη συνεδρίαση είναι προγραμματισμένη για τι Βρυξέλλες στι 5 Δεκεμβρίου 3 με 6.30 και 8 Δεκεμβρίου 9 με 12. Ευχαριστώ όλους για τη συμμετοχή τους στη σημερινή συνεδρίαση και καλό σας βράδυ. Είναι σωστό.